Συνάδελφοι, αν έχει την καλοσύνη να καθίσετε για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας, γιατί ως συνήθως ε, δυστυχώς δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Ως εκ τούτου ας ε, ξεκινήσουμε με την έγκριση της ε, ημερήσιας διάταξης και με μια διευκρίνηση που θέλω να κάνω και μια διευκρίνηση που αφορά στο σημείο υπερθμών 10. Σήμερα το πρωί είχαμε μία συζήτηση που έλαβε χώρα στην Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο κύριος Άουταλα, η κυρία Άουταλα, με συγχωρείτε, που είναι η συγγήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει στόχο ε, να προτείνει να μην συζητηθεί σήμερα το απόγευμα η δική της η έκθεση, καθότι στην Υποπιτροπή έλαβε χώρα μια διεξοδική συζήτηση. Επικράτησε, θα λέγαμε, συνένεση για το θέμα το οποίο εξετάστηκε και ως εκ τούτου ε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τροπολογίες, θα ε, αναφερθούν στον κατάλογο ψηφορίας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία το λόγο, αλλά υπάρχει πάντως αυτή η πρόταση, όπως σας είπα, να, ε, όπως σας είπα, να αναβληθεί αυτή η ε, συζήτηση. Πρόεδρος. Για... Δεν υπάρχουν γερμανικά, είπε η κυρία. Θα δούμε, λέει ο πρόεδρος. Arvoisa puheenjohtaja, juuri niin kuin te sanoitte, niin tarkoitukseni on ehdottaa, että alivaliokunnassa ei tänään käsitellä. Η κυρία Χαουτάλα. Δεν ακούγεται καλά η κυρία Ουτάλα και δεν μπορούμε να τη μεταφράσουμε. Το μικρόφωνο της δεν ακούγεται καλά. Τώρα εντάξει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έλεγα ποιες είναι οι προθέσεις μου. να συζητήσουμε αυτή την έκθεση, όχι όμως σήμερα. Και αυτό επειδή το συζητήσαμε επιμακρό στην υποπιτροπή και υπάρχει πλήρης ομοφωνία. Όμως έχουμε 117 τροπολογίες που προσπαθούν να βελτιώσουν την ε, έκθεση αυτή ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό για μένα το καλύτερο θα ήταν να αναβληθεί για την επόμενη συνάντηση της Επιτροπής αυτής. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε πως βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσε τις τροπολογίες, τουλάχιστον πολλές από αυτές, οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα πάει στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Οπότε μέχρι τότε πρέπει να το έχουμε συζητήσει και εμείς. Εάν λοιπόν συμφωνείτε, εγώ έτσι κι αλλιώς ήμουν σύμφωνος από την αρχή και ας δεχθούμε την πρόταση της κυρίας Αούταλα, ας αφήσουμε το σημείο 10 από τη σημερινή ημερησία διάταξη για κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία. Κατά πάσα πιθανότητα θα το εξετάσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Και έχω να κάνω και κάποιες ανακοινώσεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας. 14, 14 Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα ανταλλαγή απόψεων προβλέπεται με τον Όσκαρ Φενάντε Τιταράνκο που είναι ο Γενικός ε, ε, γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και είναι αρμόδιος όμως ε, για θέματα πολιτικά. Το θέμα θα είναι η πρόληψη και η διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις και η εντολή που δίδεται για την ειρήνη. Η άλλη συζήτηση στις 15 το πρωί σε νέα Στέφανο Ανίνο, Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης ΡΕΛΕΞ, ο οποίος είναι επίσης αρμόδιος για την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Και θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ε, εν ώψη της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης, ε, της Συμφωνίας γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική. Περνάμε λοιπόν στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις 23 Φεβρουαρίου και στις 8 Μαρτίου. Υπάρχουν τα ε, πρακτικά που σας έχουν κατατεθεί. Αν έχετε παρατηρήσει παρακαλώ μπορείτε να τις κάνετε. Αν όχι μπορούμε να προχωρήσουμε στην έγκριση των πρακτικών. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο σημείο που είναι η ανάγκη για στρατηγική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Κάφκασο. Ο κύριος Πόσελτ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά πρέπει να σας πω εγώ δεν μπορώ να σκέφτομαι τόσο γρήγορα. Εσείς είπατε για κάποια συνεδρίαση στις 14 ε, και στις 15 ε, Μαρτίου. Δεν θέλω, συγγνώμη, Απριλίου, Απριλίου ε, διορθώνει ο μιλητής. Και δεν θέλω βέβαια αυτό να το αμφισβητήσω. Προφανώς πρόκειται για πολύ σημαντικούς αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών. Μόνο που θέλω να πω έτσι γενικότερα το λέω, ότι αυτή η τάση που εμφανίζεται την Τετάρτη και την Πέμπτη συνεδριάσεων των πολιτικών ομάδων να προσθέτουμε και ε, συνεδριάσεις επιτροπών πριν από τις Ολομέλειες για τις οποίες πρέπει να προετοιμαστούμε και έχουμε παράλληλα και ε, συναντήσεις στην προεκλογική μας ε, περιφέρεια στην εκλογική μας περιφέρεια, διαπιστώνω όλο και περισσότερο ότι έχουμε συνεδριάσεις Τετάρτης και Πέμπτης της ομάδας, της εβδομάδας των πολιτικών ομάδων. Παλαιότερα δεν ίσχυε αυτό και πρέπει να προσέξουμε γιατί ενδέχεται κάποια στιγμή να έχουμε μόνο συνεδριάσεις και οι εκλογέ μας να μην μας έχουν δει καν στο πρόσωπο, να μην ξέρουν ότι υπάρχουμε. Εντάξει, λέει ο πρόεδρο, ε, λαμβάνουμε υπόψη μας τις ε, παρατηρήσεις σας και προφανώς ε, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντως, η συνεδρίαση που σας ανέφερα είναι την Τετάρτη το απόγευμα και η άλλη της Πέμπτης είναι το πρωί. Άρα δηλαδή δεν επικαλύπτονται με συνεδριάσεις ε, πολιτικών ομάδων. Εν πάση περιπτώσει αυτό που μας είπατε πράγματι ε, θα το λάβουμε υπόψη μας, σοβαρά υπόψη μας. Πρόεδρος, δεν καταλάβατε δεν καταλάβατε. Εγώ δεν είπα ότι επικαλύπτονται οι συνέδριασεις αυτές με τις ε, πολιτικές ομάδες, όμως επικαλύπτονται με δραστηριότητες που έχουμε στις πατρίδες μας, στις εκλογικές μας περιφέρειες. Κανονικά ήθιστε την Τετάρτη μεσημέρι να τελειώνει αυτή η εβδομάδα των πολιτικών ομάδων και μετά πάει κανείς στην εκλογική του περιφέρεια. Αυτό είναι υπεπατημένο εδώ και δεκαετίες. Και τώρα τι γίνεται. Τετάρτη και Πέμπτη όλο και προστίθενται συνεδριάσεις που σημαίνει ότι υπερκαλύπτεται η εβδομάδα εβδομάδα και δεν έχουμε αρκετό χρόνο για τους εκλογείς μας. Αυτό εννοούσα. Πρόεδρος, κοιτάξτε, στο χρονοδιάγραμμα μου είπε η γραμματεία, η πέμπτη το πρωί προβλέπεται ως ε, κανονική ημέρα για συνεδρίαση ε, συνεδριάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι με μια πεπατημένη Επίσης, με πάση περιπτώσει, αυτά που μας είπατε θα τα λάβουμε υπόψη μας ε, και θα δούμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι και εμείς ε, είμαστε υποποίηση, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Θα προσπαθήσουμε, εν πάση περιπτώσει, στο μέλλον να ικανοποιήσουμε το έτοιμά σας. Έλεγα λοιπόν ε, το σημείο 5 της ημερήσια διάταξης αφορά στην ανάγκη για στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Κάφκασο. Η συγητής είναι ο συνάδελφος κύριος Κύριλοφ και το θέμα αυτό, να σας υπενθυμίσω, ότι συζητήθηκε στην Επιτροπή μας ε, στις 27 Ιανουαρίου. Ε, επειδή όμως ε, το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό, κατετέθησαν 295 τροπολογίες, πάρα πολλές. Και ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν πολλές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον εισηγητή και τους συναδέλφους του. Επίσης η Επιτροπή για την Ενέργεια μας έστειλε μια επιστολή όπου ανα φέρεται. Η Επιτροπή παρουσιάζει αυτό το επιχείρημα, δηλαδή θέλει να μας ε, επισημάνει κάποιες ε, προτάσεις που ο εισηγητής ε, προτείνει να ενταχθούν όλες αυτές σε ένα συμβαστικό κείμενο που θέλει να μας παρουσιάσει. Χωρίς λοιπόν περαιτέρω καθυστέρηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Κύριλοφ που θα μας παρουσιάσει την εισήγησή του και τις ε, προτάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτη φορά να αναφερθώ στις κύριες ιδέες της έκθεσης. Είναι στρατηγική σημασία ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Αναγνωρίζουμε και προτείνουμε στοιχεία για τη νέα στρατηγική όσον αφορά τον Νότιο Κάφκασο. Θα ήθελα εδώ να πω ότι έχετε δίκιο για το ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την έκθεση αυτή, κάπου 300 τροπολογίες, πολλή δουλειά. Αλλά αφήστε με καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους που υπέβαλαν τροπολογίες και που συνεισέφεραν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με επικοδομητική συνεργασία στην έκθεση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές, όλους ιδιαίτερος, οι οποίοι βοήθησαν στο να συμπεριληφθούν πολλές από αυτές τις τροπολογίες μέσα σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Πετύχαμε συμφωνία για 34 συμβιβαστικές τροπολογίες, πράγμα που σημαίνει ότι έτσι καλύπτονται οι περισσότερες ε, τροπολογίες. Τώρα πέραν αυτών υπάρχουν και κάποιες τις οποίες δεν έχουμε συμπεριλάβει. Αυτό γιατί θέλουμε να παραμείνουμε ουδέτεροι και αντικειμενικοί στην έκθεσή μας. Ορισμένες από αυτές δεν βοηθούν να διατηρηθεί η ισορροπία. Ξέρετε ότι η ισορροπία έτσι καλώς είναι λεπτή. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την διαμάχη Γεωργίας-Ρωσίας ή για το Ναβόρχο Καραμπάτ. Καταλαβαίνετε ότι πολλές από αυτές τις τροπολογίες θα υποβληθούν ως προφορικές τροπολογίες. Οπότε, Έχουμε και από την Ήτρε και από την Ίντε, από την Ίντε γνωμοδότηση, από την ε, Ήτρε επιστολή. Πάντως, μαζί με τους σκιώδεις έχουμε καταλήξει σε τέσσερις ε, συμβαστικές τροπολογίες που θα συμπεριληφθούν και που απορρέουν από τις γνωμοδοτήσεις και τις επιστολές των ε, άλλων επιτροπών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο εκδημοκρατισμός, η προσέγγιση στις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά να γνωρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, που ενισχύονται μέσω στρατηγικών όπως είναι εκείνη της εταιρικής σχέσης. Συνδυάζουμε επικρίσεις, αλλά μιλάμε και για επικοδομητικά μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν θα ήθελα η έκθεση αυτή να είναι σαν μια έκθεση πρόοδου. Τώρα, να μπορώ Καραμπάχ και η Γεωργία. Είναι τα δύο προβλήματα όσον αφορά τη σταθερότητα στην περιοχή και την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Οπότε στην έκθεση Αναφέρομαι στις δύο αυτές διενέξεις και λέω ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να παίξει πιο αποφασιστική σημασία ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πόλεμο φάνηκε ότι υπάρχουν κάποιες παγωμένες διενέξεις οι οποίες παραμένουν και κάποια στιγμή ξεσπάνε και ότι άρα πρέπει να βρεθεί τρόπος να ξεπεραστούν. Δείχνει επίσης πόσο ευάλωτες είναι οι προσπάθειες που γίνονται με επενδύσεις ή με προγράμματα στην ε, περιοχή όσον αφορά την ενέργεια. Δυστυχώς, με τον ε, πόλεμο αυτό συνειδητοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να παίξει πιο ενεργό ρόλο στην περιοχή, ιδιαίτερα για να φροντίζει την πρόληψη των διενέξεων αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπιση τους. Τώρα για τον Αγώρο Καραμπάχ και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα ήταν απούσα. Απλώς στηρίζει τις διάφορες ομάδες, αλλά για μένα δεν είναι αρκετό αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει στα σοβαρά το νέο της ρόλο βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διαμεσολαβητής που τον έχουν δεχτεί και δύο πλευρές. Και γι' αυτό πιστεύω ότι όταν μιλάμε για την στρατηγική μας την περιοχή, με την έκθεσή μου θα πετύχω την στήριξη της Επιτροπής αυτής, ώστε να καταλήξουμε σε κάτι θετικό όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κυρίλοφ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον σκιώδη συγκητή του ΕΛΚ, Ιμπριτζερτζικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ Συμφωνώ με την, τον εισηγητή ότι είχαμε αγαστή συνεργασία, όχι μόνο ανάμεσα στον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές, αλλά και ανάμεσα στους σκιώδεις εισηγητές. Ως αποτέλεσμα, ε, καταφέραμε να καταλήξουμε σε σχεδόν 30 συμβαστικές τροπολογίες. Μην ξεχνάτε ότι αρχίζαμε με 300 τροπολογίες, ε, και θα ήθελα να ποτίσω φόρο τιμή στη γραμματεία. Πραγματικά τα κινήθηκε αποτελεσματικά και ταχύτατα. Ούτε εμεί θέλουμε να είναι έκθεση προόδου. Μιλάμε για, την, ε, για τον προσδιορισμό τη ενωσιακή στρατηγική για τη συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου και γι' αυτό προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τις ε, ακραίες θέσεις ε, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Θέλουμε μια κοινή στρατηγική για ολόκληρη την περιοχή, χωρίς ε, να δακτυλοδεικτούμε με μονομένα κράτη ή με μονομένες σειράξεις. Εξ ονόματος του ΕΛΚ, εγώ προσπάθησα να προσδιορίσω επακριβέστερα την πολιτική της Ένωσης για θέματα όπως το ελεύθερο εμπόριο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μας τι σημαίνει για την οικονομία, για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης, ε, η κοινή στρατηγική, η εξωτερική στρατηγική, η στρατηγική ασφάλειας, ε, τι γίνεται με τους πρόσφυγες, ε, αν δεν έχει εξασφάλιση; Δεν γίνεται να επαναπροωθούμε τους πρόσφυγες αν δεν έχουμε κατοχυρώσει την ασφάλεια στις χώρες προέλευσης τους. Επίσης, ε, πώς μπορούμε να επικουρήσουμε αυτές τις χώρες ώστε να διοργανώσουν ελεύθερες ε, εκλογές ε, και πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε εμείς το κατά πόσο υπάρχει διαφάνεια στη διεξαγωγή εκλογών. Ξαναλέω, δεν θέλουμε να ονοματίσουμε κανένα δακτυλοδεικτούμε κράτη και παρόλα αυτά οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να αναφερθούμε στην ελευθερία έκφρασης και στην ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης διότι είναι τόσο ευρύτατα τα προβλήματα στην περιοχή ούτως ώστε πρέπει να ασκήσουμε πίεση και να προστατεύσουμε και τους ακτιβιστές που υπεραμείνουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα υποβάλω προφορικές τροπολογίες, ε, κυρίως ε, τεχνικού χαρακτήρα. Ο κύριος Ουγγουριάνοφ από το ΕΛΚΑ έχει υποβάλει ε, την τροπολογία 24 σχετικά με το Euronest και την εγκαθίδρυσή του και χρησιμοποιείται μία ημερομηνία και λέμε το Μάρτιο. Μα έχει περάσει ο Μάρτιος, έχουμε φτάσει στον Απρίλιο, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, οπότε θα υποβάλω προφορική τροπολογία για να διαγράψουμε αυτή την ε, ημερομηνία. Ε, και ε, ελπίζω να με υποστηρίξουν οι συνάδελφοι. Υπάρχει κι άλλο ένα προβληματάκι για μας, το ΕΛΚΑ, για την 30, τροπολογία 30. Εδώ θα ζητήσω κατά τμήματα ψηφοφορία και συμβιβασμό για το τελευταίο τμήμα, όπου μιλάμε ε, για την ένωση του ευξήνου πόντου. Θέλουμε κατά τμήματα ε, ψηφοφορία το επισημαίνουμε ήδη, γιατί μπορεί κάποιο να θέλει να υπερψηφίσει και τα δύο τμήματα ή μόνο το τελευταίο. Ε, και τα συμφωνήσαμε και με τις πολιτικές ομάδες και υπάρχουν κάποιοι που θα υποστηρίξουν το ΕΛΚΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το λόγο η κυρία Λούνα Τσεκ, η οποία είναι σκιώδης εισηγήτρια ε, των ε, Πρασίνων. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές, αλλά και την γραμματεία που δούλεψαν σκληρά για να ετοιμαστεί η έκθεση αυτή. Θέλω επίσης εκ μέρους της ομάδας μου να στηρίξω και την πρόταση του εισηγητή όσον αφορά το κείμενο του κειμένου, αλλά και τις συμβαστικές τροπολογίες. Συμφωνώ με όσα είπαν οι συνάδελφοι πριν από μένα, ότι δηλαδή θέλουμε μια κοινή στρατηγική για ολόκληρη την περιοχή. Θέλουμε να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενισχύσει το ρόλο της στα διάφορα πεδία πάνω στα οποία θέλουμε να έχουμε σχέσεις με όλες αυτές τις χώρες. Υπάρχουν ε, παρόμοια προβλήματα και στις τρεις χώρες, είτε πρόκειται για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Υπάρχουν λίγο πολύ προβλήματα σε διαφορετικά επίπεδα μεν, αλλά και στις τρεις χώρες προσπαθούμε να αναφέρουμε κάποια θέματα χωρίς να μπούμε όμως πάντα σε λεπτομέρειες. Έπειτα το θέμα της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή καταπίεση των ανθρώπων που στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή όσον αφορά την αντιπολίτευση. ποιο είναι ο ρόλο της κοινωνία των πολιτών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των ανθρώπων που υποστηρίζουν τι ε, μειονότητε, είτε είναι ε, θηλυκτικές, είτε σεξουαλικές, είτε οτιδήποτε. Ο κύριος στόχος μας λοιπόν ήταν να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενισχύσει την δημοκρατία εκεί, την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία της έκφρασης, αλλά πώς μπορεί να παίξει και διαμεσολαβητικό ρόλο με το καλό και με το άγριο, άλλοτε με το καλό, άλλοτε με το άγριο, ώστε να στηρίξει και τους κυβερνητικούς αλλά και άλλους παράγοντες της κοινωνίας εκεί, προκειμένου να έρθουν πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αξίες και στο ευρωπαϊκό τρόπο. Ένα από τα πράγματα λοιπόν που πρέπει να πω, μου έκανε εντύπωση την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στη Γεωργία με μια αντιπροσωπεία και εξακολουθώ να βρίσκομαι υπό το κράτος της ε, εντύπωσης που μου έκαναν όλα όσα είδα εκεί και στα σύνορα με την Οσετία και αλλού. Μίλησα με ανθρώπους επιτόπου και γι' αυτό λέω ότι ο ρόλος που έχει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γεωργία, αλλά όχι μόνο, και στις άλλες χώρες είναι είτε να προλαμβάνει ε, διενέξεις, είτε αυτές είναι από αυτές που έχουν μείνει κρυφές, παγωμένες για πολύ καιρό, είτε κάτι άλλο οι άνθρωποι πρέπει να ξαναβρούν τη χαρά της ζωής. Στη Γεωργία μετά τον ε, πόλεμο κάπου 200.000 άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους και δεν είναι και τόσο μεγάλη χώρα. Λοιπόν αν τα δούμε όλα αυτά στην έκθεση καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό να υποθούν και να υπάρχουν εκεί. Τώρα θέλω να αναφερθώ σε κάποιους συμβιβασμούς που έχουμε προτείνει. Χαίρομαι που πετύχαμε συμφωνία και τη συμβαστική τροπολογία αριθμός 26. Μας απασχολεί η άνοδος στις αμυντικές δαπάνες και τις στρατιωτικές δαπάνες, γιατί δεν είναι έτσι που χαλαρώνουν οι πιέσεις και οι εντάσεις, κάθε άλλο. Ένα άλλο θέμα είναι η άρνηση του Utolsat, που είναι ένας δορυφόρος που μεταδίδει εκπομπές η απαγόρευσή του λοιπόν είναι κάτι που μας απασχολεί. Ουσιαστικά οι άνθρωποι που μιλάνε ρωσικά ή κάτι άλλο, μόνο της γεωργίας της εκβάσης μπορούν να ακούνε. Εμείς δεν θέλαμε κάτι τέτοιο, γι' αυτό και βάλαμε μια συμβαστική τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να αναφερθώ και στο σημείο 6 όπου συμφώνησα με τον εισηγητή να έχουμε το πρώτο τμήμα που μιλάει για την στρατηγική όσον αφορά τα κατεχόμενα και το υπόλοιπο θα προτείνουμε κάτι στην Ολομέλεια. Δεν το έχουμε ετοιμάσει ακόμα, άρα μόνο το πρώτο κομμάτι εδώ μετράει. Έπειτα για τους πόρους ενέργειας, το ενεργειακό ζήτημα και για αυτές τις χώρες, τις ίδιες, αλλά και όχι μόνο, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ενεργειακό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό το έχουμε συμπεριλάβει. Το κύριο ζήτημα δηλαδή είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει και να ενισχύσει αυτούς στις τρεις αυτές χώρες που θέλουν ειρήνη, δημοκρατικές διαδικασίες και σταθερές κοινωνίες που να πηγαίνουν καλά και κοινωνικά και οικολογικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα ο άδερφος Νικολάη Σκιώδης από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η ομάδα των Φιλελεύθερων στηρίζει την έκθεση αυτή. Είναι μία έκθεση που περιλαμβάνει πάρα πολλούς συμβιβασμούς, πράγμα που αποδεικνύει ότι υπήρξε τεράστια συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Οι περισσότερες τροπολογίες που διατύπωσε η ομάδα μας συμπεριλαμβάνονται στις συμβαστικές αυτές τροπολογίες. Οπότε χαιρόμαστε που υπήρξε αυτή η ίση μεταχείριση για ολόκληρη την περιοχή. Και ολόκληρη η περιοχή πρέπει να συνεργαστεί, γιατί αυτή είναι μια λύση και όσον αφορά το στρατιωτικό σκέλος και όσον αφορά την συνεργασία σε άλλους τομείς μεταξύ των χωρών αυτών. Χαιρόμαστε επίσης που οι διαπραγματεύσεις του ΜΙΣΚ για τις ε, διαπραγματεύσεις τις ειρηνευτικές προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει διπλωματική συνεργασία μεταξύ των χωρών αυτών, κάτι που είναι ιδιαίτερα θετικό στο σημερινό πολιτικό πλαίσιο στην περιοχή. Εμείς πιστεύουμε πως ήταν ορθό που επιμείναμε και στην ανθρωπιστική πτυχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον ξεχασμένο πληθυσμό της Ευρώπης. Μιλάμε για 250.000 ανθρώπους και τα κατεχόμενα μετά την ε, σύρεξη πρέπει να ξαναβρούν τη ζωή τους. Εμείς λοιπόν ε, χαιρόμαστε και για τόσο αναφέρον όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης, την ελευθερία έκφρασης και γι' αυτό και θα υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Πρώτος Αντιπρόεδρος Επιτροπής ε, μας ε, και σκιώδης συγητής της ΕΦΕΝΤΗ, ο κύριος Προβέρα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη θαυμάσια δουλειά του, πολύ καλή δουλειά και του ίδιου και της γραμματείας που τον στήριξε. Κατατέθηκαν πάρα πολλές τροπολογίες, αξιολογήσαμε επίσης και πάρα πολλές παρατηρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν πολύ σύντομα να εστιάσω την προσοχή μου σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι έχει προκύψει μια στρατηγική του Κοινοβουλίου αυτή η συνεργασία προς Ανατολάς ε, ο συνάδελφος Βιγγένινγκ είναι ένας από τους ε, βασικούς ε, προτεργάτες αυτής της ε, συνεργασίας και πέρα από την οικονομική και πολιτική συνεργασία ε, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτά τα κράτη τα οποία θα επιθυμούσαν να έχουν μια στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν αυτές τις έξι χώρες που είναι Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Γεωργία, χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται και που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Στόχος λοιπόν αυτής της συνεργασίας είναι να προωθηθούν οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός και στις έξι υποψήφιες χώρες αν θέλετε αφετέρου. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό, το θέμα είναι ότι ο στόχος εξακολουθεί να είναι να ευνοηθεί η συνεργασία ανάμεσα στις ίδιες τις χώρες. Δύσκολο αυτό γιατί βεβαίω υπάρχουν διενέξεις όπως παραδείγματος χάρη η διένεξη του Ναγκόρνο Καραμπάχ και βεβαίω και η τραγική κατάσταση της Γεωργίας. Εγώ θεωρώ ότι βασικό δικό μας έργο είναι να ευνοήσουμε την ε, άμβλυνση της διένυξης, ε, την επίλυση του προβλήματος και με τον τρόπο αυτό να μην υπάρχει η ίδια ε, ένταση και αντίθεση ανάμεσα στις χώρες οι οποίες κυρίως εμπλέκονται στην περίπτωση Ναγκόρνο Καραμπάχ που είναι η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν το να αμβληνθεί η κατάσταση, αυτό σημαίνει ότι εργάζεται κανείς και πρακτικά για την ασφάλεια. Και αυτό πάλι σημαίνει ότι είναι κανείς σε θέση να εγγυηθεί, έστω κατά κάποιον τρόπο, την επιστροφή των προσφύγων, αλλά και όλων των άλλων που έχουν διασπαρεί από τη μία την άλλη πλευρά ε, της διένεξης. Αυτό που κυρίως παίζει ρόλο είναι ότι πρέπει να προκύψει ε, μια, ένα βασικό σχέδιο. Δηλαδή η εδαφική ακαιρεότητα μιας χώρας δεν μπορεί επουδενή να τροποποιηθεί, πόσο μάλλον μέσα από μια στρατιωτική επέμβαση. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζουν τα σύνορα και ελπίζουμε ότι αυτά τα σύνορα πλέον ε, είναι οριστικά. Αυτό το αναγνωρίζει αναγωνίζουν τόσο τα Ηνωμένα Έθνη μέσα από τα ψηφίσματά τους, όπως επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική που χαράσει. Κατόπιν τούτου πρέπει να εργαζόμεθα προς αυτή την κατεύθυνση. Το άλλο που θέλω να πω είναι ο ρόλος πολύ σημαντικός που κατά την άποψή μου μπορεί να διδερματίσει η κοινωνία των πολιτών για ανθρωπιστικές παρεμβάσεις. Πρόκειται για μια στρατηγική η οποία είναι παράλληλη με την ε, πολιτική, την πραγματική πολιτική και πρέπει οπωσδήποτε να τη στηρίξουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ε, συγχαρώ και τον εισηγητή και τους ε, συνεργάτες του. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Προβέρα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπροκ. Κύριε Πρόεδρε, έχω να κάνω και εγώ κάποιες ε, παρατηρήσεις. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Κυρίλοφ για την έκθεσή του και για την προθυμία που έδειξε να εξετάσει τις ε, τροπολογίες και να καταθέσει συμβαστικέ προτάσει. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλα αυτά τα οποία ήδη ελέγχθησαν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε για την ε, εταιρική σχέση με αυτές τις χώρες και να δώσουμε έτσι μια πολυδιάστατη μορφή διαβάζοντας αυτά τα κείμενα, ίσως να μην το είδα, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι μιλάμε για τις μεμονωμένες χώρες και για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτές τις μεμονωμένες χώρες. Αλλά κατά την άποψή μου δεν μιλάμε επαρκώς για τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Ίσως λοιπόν, ε, συνάδελφε κύριε Κυρίλοφ, ε, αύριο πριν από την ψηφορία μπορείτε να πείτε κάτι από αυτό, να προσθέσετε μια πρόταση. Γιατί το πρόβλημα είναι τόσο στην ανατολική εταιρική σχέση όσο και στην ε, ε, σχέση μας με τη Μεσόγειο είναι ότι αν θέλουμε πραγματικά να σημειώσουμε επιτυχία, τότε οι οικονομικοπολιτικές σχέσεις ανάμεσα στις ίδιες τις χώρες πρέπει να ενισχυθούν. Γιατί τα ποσοστά, οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τις σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως με τις σχέσεις προς τις υπόλοιπες χώρες. Παλαιότερα όλα αυτά ε, κατευθύνονται προς τη Ρωσία, η περιοχή είχε μια άμεση σχέση με τη Ρωσία. Τώρα λοιπόν εν μέρη ε, προσπαθεί να αντικαταστήσει τη σχέση αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως δεν αρκεί για την εσωτερική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Ίσως λοιπόν αύριο στις συμβαστικές προτάσεις ε, βρείτε κάποια δυνατότητα να επισημάνετε αυτή την πραγματικότητα. Νομίζω ότι η ανατολική εταιρική σχέση είναι το σωστό εργαλείο και μπορούμε και να το στηρίξουμε οικονομικά. Αυτό το αναφέρετε και εσείς ε, στην έκθεσή σας. Μέσα από αυτήν μπορεί να υπάρξει μια ζώνη ελεύθερων ανταλλαγών και δεν θα πρέπει να αφορά μόνο το Αζερβαϊτζάν, την Αρμενία και τη Γεωργία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι να υπάρχουν και ελεύθερες ανταλλαγές ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε, όπως σας είπα, αυτή την αλένδεση των κρατών. Ευχαριστούμε κύριε Μπροκ. Το λόγο έχει ο κύριος Σβόμποντα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σύντομα να πω και εγώ κάτι. Ε, τυχαία ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε και ο κύριος ε, Μπροκ. Πριν από λίγες μόνο ημέρες ε, ήμασταν στη Γεωργία και εκεί μιλήσαμε με εκπροσώπους του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας. Και ένας εκπρόσωπος από αυτούς μας είπε ότι η περιφερειακή συνεργασία είναι μια έννοια που θέλουν να μας την επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι. Εμείς όμως πρέπει να τους πούμε ότι η περιφερειακή συνεργασία είναι μία εκ των προϋποθέσεων έτσι ώστε στο μέλλον να έχετε πρόοδο. Οικονομική, πολιτική και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι μπορούμε να βρούμε κάποια διατύπωση. Γνωρίζω ότι σήμερα ε, το να πει κανεί στους Αρμενίους και στους Αζέρους ε, ξέρετε να συνεργάζεστε, αυτό είχε παράδοξο. Αν όμως δεν υπάρχει κάποια συνεργασία η οποία να αφήνει έστω κατά μέρος, κατά κάποιον τρόπο, τον Αγκόρνο Καραμπάχ, είτε πρόκειται για θέματα μεταφορών, είτε για ελεύθερες εμπορικές συνταλλαγές, αλλά είτε και για πολιτιστικά θέματα, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι εδώ στο Κοινοβούλιο με την αντιπροσωπεία Νοτιού Καυκάσου προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε συνεργασία μέσα από τον πολιτισμό. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, δεν θα υπάρχει πρόοδος. Πρέπει να βρούμε μια διατύπωση για να πούμε ότι η περιφερειακή συνεργασία είναι καθοριστικός παράγων για να μπορέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την περιοχή, να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα αυτής της περιοχής. Αν μπορείτε κάπως να το προσθέσετε, αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον κύριο Σβόμποντα. Ε, κύριε Κύριλοφ, ε, θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ, όπως σας συνεχάρισαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να κάνετε τις ε, καταληπτικές παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συναδέρφους που πήραν το λόγο μέχρι τώρα. Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους και για τις καλές τους ιδέες. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για την τόσο αποτελεσματική βοήθεια που μου προσέφεραν. Στην αρχή όμως ξέχασα να ευχαριστήσω και ένα σωρό μη κυβερνητικέ οργανώσεις που γνωρίζοντας τα περί της έκθεσης ανέλαβαν από μόνες τους την πρωτοβουλία, ήρθαν και με βοήθησαν και μάλιστα ορισμένε προειδοποίησει ήρθαν από μη κυβερνητικέ οργανώσεις που γνωρίζουν την κατάσταση στην περιοχή. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι Πρώτα απ' όλα, όπως είπε και η κυρία Γκνουβίτς και εγώ θέλω να επιβεβαιώσω ότι θα υπάρξει επιπλέον προφορική τροπολογία. Συμφωνώ με τα όσα προτείνει, γιατί είναι σωστό, όπως ακούσαμε, ότι ήδη υπάρχει στρατηγική. Αλλά θέλω να αφαιρθώ λίγο στον κύριο Μέρα Μπροκ και σβόμποτα σε αυτά που είπαν αυτοί. Είμαι πεπισμένος για το ότι η περιφερειακή συνεργασία είναι ζωτική σημασίας τώρα. Όχι μόνο για να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για να δημιουργηθεί κλίμα σταθερότητας, προκειμένου να ενισχυθούν και επαφές μεταξύ των ανθρώπων. Από την εμπειρία που έχω εγώ από το παρελθόν, είναι μια αρχή. Και οι τι λένε. Λένε εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι με τους άλλους, με το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία. Ναι, αλλά βλέπετε, και το είπε και ο κύριος Προβέρα, ότι μιλάμε για κατεχόμενα, για της βίας. Επιμένω λοιπόν και ναι, στηρίζω όλες τις ε, τροπολογίες που μιλάνε για την περιφερειακή ανάπτυξη. Συμφωνώ με όλες αυτές και από τους πράσινους θα τις στηρίξουμε βεβαίως. Αλλά αν υπάρξουν και ακόμα ευρύτερε συμβαστικέ, θα τις στηρίξω και αυτές. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ και που πρέπει να φανεί είναι όσον αφορά τον αγώνο Καραμπάχ. Εκεί να γίνει κάτι που να περάσουμε σε επόμενο στάδιο. Μέχρι τώρα δεν βλέπουμε αποτελάσματα. Και ελευθέρωση των κατεχομένων, διάδρομος ανάμεσα στον αγώνο Καραμπάχ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία. Οι συμφωνίες είχαν σχεδόν επιτευχθεί. Δυστυχώς δεν προχώρησαν όμως. Και σε αυτό πρέπει να πιέσουμε. Γιατί είμαι πεπισμένος, απόλυτα πεπισμένος. Πέρα από την τελική λύση για το τελικό καθεστώς της περιοχής, ότι πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση της συμφωνίας. Οι δύο πρόεδροι έχουν συναντηθεί. Αν γίνει αυτό το βήμα, τότε θα μπορούμε πολύ πιο εύκολα να μιλάμε για ενισχυμένη συνεργασία. Αυτό πρέπει να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Να φροντίσουμε να αλλάξει η κατάσταση στην περιοχή. Και τα ενεργειακά και οι μεταφορές όλα είναι σημαντικά, αλλά αυτά θα ακολουθήσουν εφόσον υπάρξει σημαντική αλλαγή σε αυτό το σημείο η συνθήκη της Λισαβόνας είναι καλό που μας δίνει περισσότερες εξουσίες. Συμφωνώ με όλες τις προτάσεις πάντως και χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοδομητική βοήθεια που είχα από όλους τους συναδέρφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο. Ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλου σα ότι η ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Κυρίλοφ είναι για αύριο στι 10 και 4 και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια έχει προβλεφθεί για την δεύτερη Ολομέλεια του Μαΐου. Πάμε στο σημείο υπερθμών 6 της ημερήσιας διάταξης είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας και ο ρόλος των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής. Έχουμε την έκθεση Μπίλαν, έχουν ε, κατατεθεί 39 τροπολογίες, αρκετά περιορισμένος ο αριθμός ε, στο τροπολογίες σχέδιο γνωμοδότησης και αυτές όλες ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους σκιώδεις εισηγητές. Ε, κατέληξαν αυτοί σε συμβαστικό κείμενο. Τώρα λοιπόν ο εισηγητής θα μας ε, παρουσιάσει ε, το συμβασμό και την εισήγηση. Ψηφορία είναι για αύριο το πρωί. Ο κύριος Μπίλαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ορθά είπατε, στις 23 ε, ε, Μαρτίου λάβατε την πρώτη εκδοχή του σχεδίου από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Ενωσιακή Στρατηγική για την περιοχή της ε, Βαλτικής και της Μακροπεριφέρειας. Έχει γίνει η πρώτη λοιπόν ανταλλαγή απόψεων για το κείμενο, 39 τροπολογίες. υπάρχουν ε, έχουμε συζητήσει με τους ε, σκιώδεις εισηγητές από όλες τις πολιτικές ομάδες ε, και καταφέραμε να υποβάλουμε τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες που λαμβάνουν υπόψη την πλειοψηφία ε, των ε, τροπολογιών που είχαν υποβληθεί σε εκείνη τη συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιότητες εισηγητές από όλες τις πολιτικές ομάδες και όπως είπατε πρόεδρε, αύριο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία και αναμένω τις ε, τελικές παρατηρήσεις από πλευρά των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφος Κίλαμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κέλαμ. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία και καταφέραμε ε, να καταλήξουμε σε συνένεση, όλες οι πολιτικές ομάδες να καταλήξουν σε συνένεση για τις συμβαστικές τροπολογίες. Τέσσερις είναι ικανοποιητικές για το ΕΛΚ. Το βασικό πρόβλημα με αυτήν την γνωμοδότηση ήταν ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πρέπει να εκδώσει δική της γνωμοδότηση για στρατηγική της ε, ε, Βαλτικής θάλασσας που κανονικά συνιστά εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάτε ότι η βόρεια διάσταση, η πρώην βόρεια διάσταση σχετίζεται με εξωτερικές ε, σχέσεις. Φυσικά όμως η έκθεση του κυρίου Μπίλαν πρέπει να καλύπτει και τις εξωτερικές πτυχές της πολιτικής. Καταφέραμε να αποφύγουμε ένα κίνδυνο από, στην πρώτη εκδοχή. Λέγαμε ότι ε, το κατά πόσο θα είναι επιτυχή στρατηγική για τη Βαλτική συνδέεται με την, ε, τις εξωτερικές ε, είναι συνάρτηση μάλλον των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τώρα πλέον καταργήσαμε αυτή Τη τη φράση και λέμε συμβαστική τροπολογία ότι θα ήταν καλύτερο αν είχαμε επικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους. Ε, μας ικανοποιεί ε, αυτή η διατύπωση, αυτή η νέα διατύπωση. Καταλήξαμε και σε μια ικανοποιητική συμβαστική τροπολογία για τις σχέσεις με την Ρωσία ε, σε ένα επικοδομητικό κατά τη γνώμη μου πνεύμα. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως ε, στην τροπολογία επαριθμών 4 που σχετίζεται με την ε, χρηματοδότηση της ε, στρατηγικής για τη Βαλτική. Προέκυψε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη προσανατολιζόταν προς το πνεύμα που διέπει την βόρεια διάσταση. Άρα τα 20 εκατομμύρια ευρώ που είχαν εξασφαλιστεί για τη στρατηγική ή για τη Βαλτική μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, για τη φετινή χρονιά μόνο για τις εξωτερικές σχέσεις. Και η τροπολογία 4 προτείνει διόρθωση για το προϋπολογισμό του 2011. Ως προς τις άλλες ε, τροπολογίες, ε, το ΕΛΚ συζήτησε τις τροπολογίες 25 και 26 και συμφωνήσαμε με αυτές στο μέτρο που και οι λοιποί θα συμφωνήσουν με το συμβαστικό μας κείμενο που καταρρεί την αιρεσιμότητα. Μόνο έτσι το ΕΛΚ θα μπορέσει να υποστηρίξει τις τροπολογίες 25 και 26. Κατόπιν θα υποβάλουμε και προφορικές τροπολογίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε στην Άλφος Μίρσκι. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία που είχαμε. Ε, είμαι ο σκιώδης εισηγητής ε, των σοσιαλιστών ε, και εξ ονόματος ομάδας μου θα επιστήσω την προσοχή σας σε τρεις τροπολογίες, 24 έως και 26. Προτείνω να καταψηφιστούν αυτές οι τροπολογίες. Υπευλήθησαν από τον εισηγητή και από τους συναδέλφους του της ιδίας πολιτικής ομάδας αλλά δεν είναι καθόλου λογικές ούτε και εξυπηρετούν τον ε, επιδιωκόμενο με την έκθεση στόχο. Ε, διότι μιλάμε για το πρόγραμμα για τον Nord Stream, τον αγώνα Nord Stream, που έχει σοβαρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επίσης αναφερόμαστε στις κοινέ στρατηγικές ασκήσεις ε, της Ρωσίας και της Λευκορωσίας που συνδέονται με αυτό το πρόγραμμα. Μα από πού αντιλείται αυτές τις πληροφορίες. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια φήμη μόνο. Ίσως βέβαια έχετε πηγές που δεν γνωρίζω. Ενημερώστε με παρακαλώ. Σας υπενθυμίζω ότι οφείλουμε να επαληθεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία και μόνο τότε μπορούμε να τις συμπεριλαμβάνουμε τις πληροφορίες ε, ε, στα σχέδια. Ε, κρίνω ότι είναι περιττές αυτές οι πληροφορίες διότι τα κράτη της Ένωσης έχουν ήδη συμφωνήσει για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Ευχαριστούμε κύριε Μίσχη, κύριε Πρόεδρος. Ο κύριος Γιάτε Μάκη τώρα. Thank you, Mr. President. I would also... Η κυρία Γιατεμάκη, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους τους σκιώδεις για την πολύ καλή συνεργασία μας, χάρη στην οποία καταλήξαμε σε ε, συνένεση και συντάξαμε τις συμβαστικές ε, τροπολογίες και ευελπιστώ να ικανοποιούν αυτές όλους τους ε, συναδέλφους. Θα τονίσω ότι δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω γραφειοκρατικές δομές. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρακτική συνεργασία και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Θα ήθελα να τονίσω όλους ιδιαίτερος την ε, συνεργασία σε, για περιβαλλοντικά ζητήματα θέμα που συζητήθηκε και ελπίζουμε πραγματικά να εμπλακεί με πιο ενεργό τρόπο η Ρωσία σε αυτή τη συνεργασία. Παρόλα αυτά, κλείνω λέγοντας, τους όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε κυρία Γιατεμάκη. Ο κύριος Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο δικός μας ο σκιώδης ηγητής είναι ο κύριος Ταραντ, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να έρθει, γι' αυτό θα μιλήσω εγώ εκ μέρους του. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή και θα ήθελα κυρίως ε, να επισημάνω ότι κατά τη δική μας άποψη οι τροπολογίες ε, μπορούν να εγκριθούν και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα αναφερόμενος ε, σε αυτά που είπαν ε, οι συνάδελφοι να πω και εγώ κάτι για τις τροπολογίες 24, 25, 26. Ίσως ε, Πολλοί από εσάς να πιστεύουν ότι εγώ δεν δέχομαι αυτόματα όλες τις τροπολογίες αυτής της ε, πολιτικής ομάδας, αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτές οι τροπολογίες είναι αντιρωσικές. Η τροπολογία υπερθμών 25 εκφράζει την ανησυχία, παραδείγματο χάρη, για την εφαρμογή του ε, αγωγού North Stream και κατόπιν γίνεται κάποια διευκρίνηση με την έννοια ότι γίνεται ιδιαίτερη μνήμα των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Εγώ λοιπόν πιστεύω ανεπιφύλακτα ότι εδώ έχετε ε, δίκιο στην αδελφέ ότι το πρόγραμμα, το σχέδιο αυτό έχει ήδη εγκριθεί. Παρόλα αυτά όμως είναι απολύτως απαραίτητο να ασχοληθούμε με τα περιβαλλοντικά. Και γι' αυτό λοιπόν ότι εγώ θέλω να πω αυτή, τον το εκφράζουμε εγώ το κρίνω ως ε, εχθρικό προς τη Ρωσία, αντιρωσικό. Κατά την άποψή μου, το 24, εγώ δεν το κρίνω με τον ίδιο τρόπο. Και αν ισχύουν αυτά που αναφέρονται στο 24, 25, 26 και κάτι τέτοιο πρέπει να διευκρινιστεί μέχρι την ε, ψηφοφορία, δεν καταλαβαίνω γιατί ε, το να διαπιστώνει κανείς κάτι απλά και μόνο αυτομάτως πρέπει να οδηγεί ε, τους άλλους να πιστεύουν ότι είναι εχθρός της Ρωσίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Πιτικόφα ε, Αλέτσκι. Παλέκης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις, ε, διότι κρίνω ότι ε, πρότειναν, υπέβαλαν λογικές ε, τροπολογίες και θα ήθελα να αναφερθώ στην μεγάλη σημασία του Καλίνιγκραντ ε, οφείλουμε να τονώσουμε την ε, κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή αυτή, γιατί είναι μια πύλη και, ε, και αυτό ταυτόχρονα για τη συνεργασία της Ευρώπης με τη Ρωσία και μπορεί να λειτουργήσει η περιοχή ως βαρόμετρο των σχέσεων της Ένωσης με τη Ρωσία και ένα βαρόμετρο επίσης των ηγετικών προθέσεων της Μόσχας. Ε, θα μας βοηθούσε να αξιολογήσουμε την υλοποίηση της στρατηγικής ε, για την περιοχή αυτή σε σχέση με την ε, στρατηγική της Ένωσης για το 2020. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να... και θα υποβάλουμε προφορική τροπολογία για αυτό το θέμα. La parola al collega Svoboda. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Svoboda έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα του North Stream. Εγώ προσωπικά είμαι ε, κατηγορηματικός ε, υποστηρικτής ε, του Ναμπούκο, του ανταγωνιστικού αγωγού. Ε, κάποιοι βέβαια συνάδελφοι ε, κέρδισαν και γι' αυτό δεν θεωρώ ότι έχει νόημα να μιλάμε συνέχεια για το North Stream. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα κατά πόσον κάποιο είναι φίλο ή αντιρωσικό. Αυτά για μένα δεν είναι κριτήρια που παίζουν ρόλο. Όμως αν τελικά η πρώτη τροπολογία λέει ότι Κατά την εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη τα περιβαλλοντικά ε, στοιχεία. Εδώ ο κύριος Μπιουτικόφε έχει δίκιο. Σωστό αυτό το επιχείρημα και εγώ τάσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ της διαφάνειας των πραγμάτων. Όχι όμως με μια ε, διατύπωση περικοκλάδα. Εγώ θέλω να πω με απόλυτη σαφήνεια ότι αν τελικά πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα, μα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα περιβαλλοντικά θέματα. Σωστό αυτό. Δεύτερον, ερχόμεθα εδώ σε αυτά τα θέματα των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων. Εγώ ε, δεν θέλω που δεν είναι στρατιωτικές κοινέ ασκήσει με τη Λευκορωσία. Αλλά τι έγινε τελικά. Είπαν ότι θέλουμε να περασπιστούμε τις ανατολικές περιοχές ή όχι. Αν το είπαν είναι χαζό. Αν δεν το είπαν τότε και εμεί τι το ξαναλέμε και το λέμε. Αυτό το allegedly στα αγγλικά, είναι σαν να τους λέμε ότι, ξέρετε, δεν το ξέρουμε και ακριβώς, αλλά θέλουμε να σας κατηγορήσουμε. Δεν βρίσκουμε βέβαια λόγο να σας κατηγορήσουμε, αλλά βάζουμε αυτό το allegedly στα αγγλικά. Κατά κάποιον τρόπο δημιουργούμε δυσπιστία, αλλά χωρίς λόγο. Αν υπάρχουν ε, ε, αποχρόντες λόγοι, τότε πράγματι να ασκήσουμε ε, κριτική. Αλλά τώρα δεν έχει νόημα να λέμε ότι υπάρχει κίνδυνος κάποιος με βόμβα να ε, ανατινάξει το North Stream. Αυτές, ξέρετε, είναι διατυπώσεις οι οποίες προκαλούν δυσπιστία, χωρίς να εκφραζόμεθα με σαφήνεια. Και τι γίνεται τελικά, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Μία καλή έκθεση επιδεινώνεται. Κακό αυτό. Ο συνάδελφος κύριος Μπροκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, οι δύο τελευταίες ε, παρεμβάσεις με ενεθάρρυναν να πω και εγώ λίγα λόγια. Αναμφισβήτητα λοιπόν τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμφωνούν όλοι είναι ότι πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη τα θέματα του περιβάλλοντος. Οφείλουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε μία διαφοροποίηση. Υπάρχουν τα τυπικά ε, και η Φινλανδία, Δανία, Γερμανία προφανώς επιβεβαιώνουν αυτές τις ε, διαπιστώσεις, τις τυπικές. Το δεύτερο είναι ότι παρόλα αυτά πρέπει κανείς να μεριμνήσει ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις. Και τρίτον, γίνεται λόγος για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 8 Ιουλίου 2008. Ίσως μπορούμε να πάρουμε την διατύπωση του κυρίου Σβόμποντα και να πούμε ότι καλούμε και την Επιτροπή να μας ε, ενημερώσει κατά πόσον σύμφωνα με το έτοιμά μας της 8 Ιουλίου 2008 τηρήθηκαν οι πολιτικές ε, προϋποθέσεις. Νομίζω ότι το συζήτησαμε αυτό στην πολιτική ομάδα. Και αν γίνει, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και κατόπιν τούτου, δεν θα μιλάμε έτσι γενικά, δεν θα εκφράζουμε ανησυχία για την εφαρμογή, απλά ε, θα προβάλλουμε αυτό το θέμα και θα παρακαλέσουμε την Κομισιό να το εξετάσει για να δούμε κατά πόσον τηρήθηκε. Το δεύτερο που θέλω να πω πράγματι έχει σχέση με τις ε, στρατιωτικές ασκήσεις. Ένα πράγμα είναι σαφές και αυτό το επισήμανε ο ΑΣΕ, ότι η άσκηση αυτή έλαβε χώρα στην Οσετία. Είχε ε, προκηρυχθεί, είχε ανακοινωθεί, άρα δηλαδή τηρήθηκαν όλες οι τυπικές ε, προϋποθέσεις ε, ε, που πρέπει να τηρούνται για τις ασκήσεις. Το ότι δεν μας αρέσει αυτό είναι άλλο θέμα. Μόνο που όταν τηρούνται τυπικά οι προϋποθέσεις πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί και εμείς επιθυμούμε να έχουμε ας πούμε κοινέ ασκήσεις του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία. Και δεν μπορούν εκεί να παρέμβουν οι Ρώσοι και να πούνε δεν σας το επιτρέπουμε, αν τυπικά είμαστε εντάξει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ισχύει και για τις δύο πλευρές, έτσι ώστε καμία από τις δύο πλευρές να μην διεκδικεί ζώνη δικής της επιρροής. Τώρα, αυτό το allegedly, αυτό ε, που είπε ο σταρφος κύριος Σβόμποτα και διαφωνεί. Ίσως μπορούμε να προσπαθήσουμε, όπως είπε και ο συνάδελφος κ. Πιουτικόφα, να το επανεξετάσουμε το θέμα, το ε, κατά πόσον ε, πράγματι υπάρχουν ε, στόχοι και καθήκοντα στην άσκηση αυτή. Αν ισχύει, τότε πράγματι θα πρέπει να πάρουμε το θέμα σοβαρά. Ότι δηλαδή η Ρωσία προστατεύει με τη Λευκορωσία ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν το βρίσκω και ιδιαίτερα αστείο, αυτό μπορούμε να το πούμε. Όμως θα πρέπει να έχουμε αποδείξεις για αυτό το θέμα. Ε, να μην είναι ένας ισχυρισμός και ίσως ο εισηγητής ε, μέχρι την ψηφοφορία μπορεί να μας καταδείξει το δρόμο για να καταλήξουμε σε μια συμβαστική πρόταση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μπροκ. Το λόγο έχει τώρα ο στάλφος κύριος Λαντσμπέργκης. Ευχαριστώ. Αναρωτιέμαι αυτά που λέμε για την τροπολογία 25. Μα υπενθυμίζουμε εδώ το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2008 με μεγάλη πλειοψηφία. Και τώρα λέμε ότι είναι αντιρωσικό το να υπενθυμίζουμε το ψήφισμα. ολόκληρο το ψήφισμα ήταν αντιρωσικό. <laughs> Κατηγορήθηκε το κοινοβούλιο ολόκληρο ότι ήταν ε, ε, κατά της Ρωσίας. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα λέμε αυτά. Εγώ θυμάμαι ότι τότε διάφορες ε, που προώθησε η Γκασπρόμ όντως δεν εγκρίθηκαν. Ε, μα τι, τόσο τραγικό είναι αυτό. Ε, για να καταφερόμεθα κατά αυτόν τον τρόπο κατά ενός ε, ψηφίσματος του Κοινοβουλίου. Αν ε, σε κάποιον δεν αρέσουν τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, εντάξει, αλλά δεν είναι λόγος αυτός. Το λόγο Σίβιετς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι εδώ μιλάμε για μία έκθεση. Είναι μια έκθεση η οποία επεξεργάζεται ένα θέμα το οποίο ίσως να μην είναι το πιο σημαντικό θέμα που εξετάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι και περιθωριακή έκθεση. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι για ένα θέμα κλειδί. Είναι εξάλλου η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που είναι η αρμόδια επί της ουσίας κοινοβουλευτική επιτροπή για αυτή την έκθεση. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή, η Περιφερειακή Επιτροπή, είναι εκείνη η οποία θα δώσει τελικά το στήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμάς μας ζήτησαν να γνωμοδοτήσουμε. Εννοείται ότι κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, έρχονται διάφορες προτάσεις. Θέλουμε να σώσουμε τον κόσμο, θέλουμε να φτιάξουμε ένα νέο αγωγό φυσικού αερίου, θέλουμε να βάλουμε, να βγάλουμε στρατιωτικές δυνάμεις. Εγώ νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό τελικά ξεχνάμε ποιος είναι ο δικός μας ο ρόλος που είναι να γνωμοδοτήσουμε στην έκθεση αυτή. Η Επιτροπή Εξωτερικών ε, Υποθέσεων μιλάει πάρα πολλές φορές για τη συνεργασία μας με την Ρωσία. Μιλάμε πολύ για την ασφάλεια, για την ασφάλεια στην περιοχή της Βαλτικής και νομίζω ότι όταν αναφερόμαστε σε αυτή την έκθεση και όταν θέλουμε να προτείνουμε μεγάλες αλλαγές, αυτό δεν είναι επικοδομητικό. Γιατί ακόμα κι αν υπερψηφιστούν τέτοιες προτάσεις, παραμένουν περιθωριακές σε σχέση με το κύριο ζήτημα που εξετάζει η έκθεση αυτή. Μας ζητήθηκε να γνωμοδοτήσουμε πάνω στην έκθεση που υποβάλλει η Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό πρέπει να κάνουμε, σε αυτόν επικεντρωθούμε. Αλλιώς ξεφεύγουμε και δίνουμε την εντύπωση ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε τη μεγάλη πολιτική με μια τροπολογία που τελικά είναι πολύ μικρή σε σχέση με ολόκληρη την έκθεση. Όσο πιο σύντομη είναι η γνωμοδότησή μας, τόσο το καλύτερο. Επιπλέον να προσθέσω και κάτι ακόμα. Όταν ακούω όλα όσα λέγονται για τους στρατιωτικούς ελιγμούς, κανένας δεν θέλει στρατιωτικούς ελιγμούς ε, στα σύνορα. Ούτε και μένα με ικανοποιεί κάτι τέτοιο, μια τέτοια κατάσταση. Όταν ακούω ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία θέλουν μαζί να στηρίξουν τον αγωγό που φτιάχνουν μαζί η Γερμανία και η Ρωσία, ε, τελικά ποιο θέλει να τα βάλει με αυτόν τον αγωγό, αφού τον φτιάχνει η Ρωσία από τη μια μερία και από την άλλη μια, μια χώρα του ΝΑΤΟ. Conclude, conclude Τελευταίος ε, συνάδελφος Βιγενή και τελειώνει η παρεμβάση. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος γιατί λίγο πολλοί συνάδελφοι είπαν αυτά που είχα να πω κι εγώ. Να προσθέσω όμως ότι σε μια τέτοια γνωμοδότηση πρέπει να έχουμε συνένεση όσον αφορά το θέμα αυτή τη φορά τη Βαλτική. Εμείς όμως τελικά οδηγούμεθα σε αντιφατικές τροπολογίες, οπότε σε μια κατάσταση που σίγουρα δεν είναι βιώσιμη. Δεν θα καταλήξει πουθενά. Κυρίως αυτό ισχύει για τις τροπολογίες 25 και 26. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος είναι υπέρ ή κατά της Ρωσίας. Το θέμα είναι το ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια γνωμοδότηση ε, όπου πρέπει να περιλαμβάνονται θέματα τα οποία έχουν να κάνουν άμεσα με την ε, σχετική έκθεση και όχι με άλλα. Οπότε, προσοχή στη διατύπωση της 25 και κυρίως της 26 που έχει να κάνει με θέματα τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ το θέμα της γνωμοδότησής μας. Και εξάλλου, μάλλον θα απορρευθούν, αλλά και αν δεν απορρευθούν και εγκριθούν, θα έχουμε τεράστιες δυσκολίες στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστούμε το στόχο για τις ε, τελικές παρατηρήσεις και σχόλιο ο συνάδελφος κ. Μπίλαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε διστάμενες απόψεις ε, και διαπιστώνουμε όλοι ότι υπάρχει χάσμα ανάμεσα στις απόψεις των μεν και των δε. Γι' αυτό και σας είπα στην αρχή ότι χαίρομαι που καταφέραμε παρόλα αυτά να καταλήξουμε σε τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες όπου συμπεριλάβαμε το περιεχόμενο της πλειοψηφίας των αρχικών 39 τροπολογιών. για τις τροπολογίες, ε, για τον Nord Stream, ή ε, την ε, στρατικοποίηση κτλ. Δεν είχα εγώ συμπεριλάβει αρχικά τα ζητήματα αυτά στις συμβαστικές τροπολογίες. Πλην όμως θεωρώ ότι έχουμε το δικαίωμα στην πολιτική μου ομάδα να υποβάλουμε τέτοιες τροπολογίες. Ο κύριος Μίσκι μας μίλησε για την τροπολογία 25, αλλά νομίζω ότι το απάντησαν ε, πολλοί βουλευτές. Ευχαριστώ τον κύριο Λαντσπέρκης και τον εκπρόσωπο της ομάδας των Πρασίνων. Όντως, ε, μνημονεύεται σε αυτή την τροπολογία ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στην προηγούμενη θητεία. Δεν ήσασταν τότε βουλευτές κύριε Μίσκη, και ίσως δεν το γνωρίζατε. Ε, για την προφορική τροπολογία τώρα που υπέβαλε ο κύριος Κέιλαμ εξ ονόματος του ΕΛΚ, η δική μου πολιτική ομάδα απαντά ότι ναι, μπορούμε να εγκρίνουμε αυτήν την προφορική τροπολογία σας. Για την ε, τροπολογία 26 και όλες παρατηρήσεις, ε, που σχετίζονται με αυτήν και που υπέβαλε ο κύριος Μπρόκ. Κοιτάξτε, η προφορική τροπολογία του ΕΛΚ είναι λογική και την εγκρίνουμε. Νομίζω πριν τελική ψηφοφορία θα καταλήξουμε σε συνένεση. Ε, για τις παρατηρήσεις του κυρίου Σίβιτς, αν θεωρεί ότι το ζήτημα του Nord Stream δεν πρέπει να αναφερθεί πουθενά, να ε, απευθυνθείτε στον κύριο Λένιτζακ από τη δική σας ομάδα. Εκείνος ε, ανέφερε στην έκθεσή του το θέμα του Nord Stream. Ε, για την τροπολογία 26 πάλι το ίδιο ζήτημα για τις στρατιωτικές ασκήσεις, ασκήσεις συγγνώμη, της, η Ρωσία δεν δέχτηκε ότι ο στόχος ήταν η υπεράσπιση του αγωγού Nord Stream, αλλά πρόκειται για στρατικοποίηση της περιοχής ε, της Βαλτικής. Ε, αυτό εντάσσεται στη λογική ε, του ψηφίσματός μας εκεί εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης, εισηγητές. Ε, είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση ε, και ευελπιστώ να υπερψηφίσουν όλοι οι συνάδελφοι το σχέδιο. Πολύ ωραία λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή τον κύριο Μπίλαν και να πω κάτι που είναι γνωστό στις 8 Απριλίου, αύριο δηλαδή ε, θα ψηφιστεί η έκθεση εδώ στην Επιτροπή και στις 27 θα συμβεί ακριβώς ε, το ίδιο στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Ε, θα ήθελα ο συνάδελφος Κόβακ να κάτσει δίπλα μου και να δεχθούμε τον επόμενο εισηγητή, τον κύριο Μιγκαρέλη. Θα, από κοινού θα έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με την ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Είναι μια δική μας επιτροπή η οποία συνεδριάζει από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας της οποίας ε, προεδρεύει ο συνάδελφος κ. Κόβαλ. Ας ε, καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Μιγκαρέλη, ο οποίος είναι αναπληρωτής γενικό Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Υποθέσεων και πλέον είναι συχνά φιλοξενούμενος στη δική μας την Επιτροπή. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το σημερινό θέμα αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία εν ώψη της Συμφωνίας Σύνδεψης, ε, διαπραγματεύσεις υπό τον κύριο Μουγκαρέλη, άρα δηλαδή πλέον πλέον αρμόδιος για να με ενημερώσει για τις εξελίξεις και για να απαντήσει στις ερωτήσεις μας όσον αφορά το θέμα αυτό είναι ο κύριος Μουγκαρέλη. Επίσης ε, είμαστε όλοι λιγάκι περίεργοι ε, και θέλουμε να μας απαντήσει σχετικά με το πότε πιστεύει ότι θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, οι διαπραγματεύσει που τρέχουν δηλαδή, η δική μας Επιτροπή αποφάσισε να ορίσει έναν εισηγητή, ε, τον κύριο Λεγκούτκο, που έχει ως ε, εντολή εκ μέρου μα να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών των διαπραγματεύσεων και βεβαίως θα έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει. Το Κοινοβούλιο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το 2007 ενέκρινε ένα κείμενο στο οποίο ορίζεται, καθορίζεται η δική μας η θέση σχετικά με την εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή. Και μετά από όλα αυτά νομίζω ότι ήρθε πλέον η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε το ρόλο στον εισηγητή μας, τον κύριο Μιγκαρέλη, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να παρέμβει. Ευχαριστώ. Έχω για άλλη μια φορά την ευκαιρία να σας μιλήσω για τις πραγματεύσεις όσον αφορά την συμφωνία με την Ουκρανία. Πριν σας πω πού ακριβώς βρισκόμαστε μετά από την τελευταία συνάντηση που είχαμε, πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος Γιαννούκοβιτς που πρόσφατα εξελέγει πήγε στις Βρυξέλλες. Ήρθε την 1η Μαρτίου εδώ και ε, μίλησε πολύ καθησυχαστικά όσον αφορά τον προσανατολισμό της χώρας του υπέρ της Ευρώπης μετά από διάφορα που ακούστηκαν στην προεκλογική εκστρατεία, είπε ξεκάθαρα ότι οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσανατολισμός της χώρας, όπως επίσης και συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Άρα, η κατάληξη της συμφωνίας θα προχωρήσει γρήγορα. Όπως σας έχω ήδη πει, οι διαπραγματεύσεις για την νέα αυτή συμφωνία ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2007. Αυτό σημαίνει ότι εδώ και τρία χρόνια περίπου είμαστε σε διαπραγματεύσεις έντονες και ένα χρόνο μετά την ένταξη των διαπραγματεύσεων, τον Απρίλιο δηλαδή του 2008, μετά από την ένταξη στον ΠΟΕ της Ουκρανίας, μπορέσαμε και ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις και για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, πλήρης και σε βάθος. Αυτό σημαίνει Πέρα από τους ε, δασμούς που καταργούνται, προβλέψαμε επίσης και άλλα πράγματα, όπως την άρση όλων των μη δασμολογικών ε, εμποδίων. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν από το 2007 προχωράνε μέσα σε ένα πνεύμα ενθουσιασμού από πλευρά των Ουκρανών εταίρων μας, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το 2009 στην προεκλογική εκστρατεία ε, επιβραδύθηκαν κάπω οι διαπραγματεύσει κάτι το οποίο δεν εκπλήσει κανέναν. Αυτό φάνηκε από τις διαπραγματεύσει που είχαμε για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, γιατί ήδη τότε φάνηκε ότι ότι υπήρχαν κάποια συμφέροντα τα οποία οδήγησαν τους διαπραγματευτές από πλευρά της Ουκρανίας να επιβραδύνουν τους ρυθμούς των διαπραγματεύσεων. Έχουμε κλείσει προσωρινά 30 κεφάλαια, τα οποία θα μας επιτρέψουν να πιέσουμε την Ουκρανία προς ε, ρυθμιστικά πλαίσια που αντιστοιχούν με αυτά που έχει η Ευρώπη σε διάφορους τομείς, όπως είναι η γεωργία, το περιβάλλον, οι μεταφορές, τα στατιστικά δεδομένα και τα τελωνία το προήμιο οι στόχοι και οι κύριες αρχές έχουν ολοκληρωθεί προσωρινά. Για το θέμα πολιτικός διάλογος μπορέσαμε και συμφωνήσαμε όσον αφορά τη θεσμική δομή για να συνεχιστεί ο πολιτικός διάλογος. Για το διάλογο και τη συνεργασία όταν πρόκειται για την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα στην Ανατολική Ευρώπη έχουμε προχωρήσει για την πρόληψη των ε, σειράξεων, των κρίσεων, για την συνεργασία, την τεχνική και τη στρατιωτική, για την καταπολέμηση της διάδοσης εξοπλισμού μαζικής καταστροφής, για τον αφοπλισμό και τον έλεγχο των όπλων, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τώρα, στον πολιτικό διάλογο Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Το πρώτο είναι βέβαια το αίτημα της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο είναι το αίτημα της Ουκρανίας για να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία σύντομα. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το παρόν γι' αυτό είναι να προβλέψει ένα καθεστώς χωρίς θεώρηση, αλλά μακροπρόθεσμα και υπάρχουν επίσης και συζητήσεις όσον αφορά τη διατύπωση στην οποία θα καταλήξουμε για τις αρχές που έχουν να κάνουν ε, με την εδαφική ακαιρεότητα και την κυριότητα της χώρας αυτής. Αυτό όσον αφορά τον πολιτικό διάλογο. Για την δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια τώρα, μπορέσαμε και συμφωνήσαμε για το θέμα του κράτους δικαίου, την τήρηση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για την συνεργασία στο θέμα της μετανάστευσης, του ασύλου και των θεωρήσεων, για το θέμα της διαχείρισης των συνόρων, την μετακίνηση ατόμων, την νομιμοποίηση παράνομου χρήματο, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ε, καταπολέμηση παντός είδους ε, λαθρεμπορίου, ναρκωτικών μεταξύ άλλων, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και διαφθορά. Επίσης, συνεχίζονται διαπραγματεύσεις στον τομέα απασχόλησης των παράνομων μεταναστών, την μετακίνηση ατόμων, τους κανόνες υποδοχής και την δικαστική συνεργασία στο τομέα του αστικού δικαίου. Όσον αφορά την οικονομική συνεργασία και την συνεργασία ανατομής, έχουμε ολοκληρώσει σε 30 τομείς προσωρινά τις διαπραγματεύσεις, κάτι το οποίο θα επιτρέψει στην Ουκρανία για άλλη μια φορά να ε, βρεθεί στα κοινοτικά πρότυπα και προδιαγραφές για να διαχειριστεί διάφορα θέματα σε αυτούς τους 30 τομείς. Δεν θα σας τους απαριθμίσω τώρα για να μην σας κουράσω, αλλά εφόσον θέλετε τις έχω τις λεπτομέρειες και ευχαρίστως να σας τις πω. Στον εμπορικό τομέα τώρα, όπως ε, σας είπα εδώ και δύο χρόνια έχουμε διαπραγματευτεί μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών πλήρη και σε βάθος μπορέσαμε ήδη να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις για τους δασμούς υπηρεσίε, υπηρεσίες, επενδύσεις, ανταγωνισμό, ε, φόρο ανάπτυξη και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για 14 κεφάλαια, ε, τρία προσωρινά έχουν κλείσει που έχουν να κάνουν ε, με την προέλευση, την συνεργασία στα τελωνία και τη διευκόλυνση του εμπορίου, όπως επίσης και για τους κανόνες που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια. Εννοείται ότι οι συζητήσεις έχουν να κάνουν με τους κανόνες σε τομείς που έχουν να κάνουν με την υγιεινή, την, ε, την ιατρική, όπως επίσης και με τους τεχνικούς δεσμούς στις ε, συναλλαγές μας. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε πιο έντονα τους επόμενους μήνες. Τώρα πότε ακριβώς οι διαπραγματεύσεις αυτές θα ολοκληρωθούν είναι δύσκολο να το πω. Εφόσον από πλευράς της Ουκρανίας κάνουν όπως κάνανε και τα τρία προηγούμενα χρόνια, δηλαδή με έντονου ρυθμούς να προχωρήσουν, θα μπορέσουμε μέσα στους επόμενους 12 μήνες να κλείσουμε τις διαπραγματεύσει. Για το πολιτικό σκέλος πιο γρήγορα. Για το εμπορικό σκέλος που είναι πιο τεχνικό θα μας χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της Κομισιόν, 6 με 12 μήνες μας χρειάζονται. Και πάλι, επαναλαμβάνω, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση από πλευρά της Ουκρανίας. Έτσι λοιπόν συνοψίζω την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Για να ολοκληρώσω, Θέλω να προσθέσω ότι έχουμε φροντίσει για διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στη Νέα Συμφωνία πριν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις. Και γι' αυτό έχουμε συμπεριλάβει μία ατζέντα σύνδεσης εδώ και λίγο καιρό που αντικαθιστά το πρόγραμμα δράσης το οποίο είχαμε καταλήξει όσον αφορά την πολιτική καλής γετνίασης πριν από τέσσερα χρόνια. Και χάρη στην εφαρμογή λοιπόν αυτής της ατζέντα για τη σύνδεση μπορούμε ήδη από τώρα να θέσουμε σε εφαρμογή κάποιους προσανατολισμούς οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην συμφωνία αυτή που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί όπως είπαμε. Επαναλαμβάνω ότι εφόσον η πολιτική βούληση υπάρχει από πλευρά της Ουκρανίας σε λίγους μήνες θα έχουμε ολοκληρώσει τι διαπραγματεύσει και γι' αυτό αποφασίσαμε ήδη να θέσουμε σε εφαρμογή την ατζέντα για την οποία σα μίλησα μόλι τώρα. Ευχαριστούμε, ο συνάδελφος Κόελ έχει το λόγο που είναι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν πολλά θέματα που αξίζει τον κόπο να συζητήσει κανείς και να υπογραμμίσει. Έχω λοιπόν ερωτήσεις για διάφορες πτυχές και πάνω απ' όλα όσον αφορά το πλαίσιο της τελευταίας μικτής συνάντησης που είχε η Επιτροπή. Έχω την αίσθηση ότι ο Επίτροπος όταν πρόκειται για το καθεστώς χωρίς ε, θεωρήσεις είχε μια διαφορετική άποψη από αυτήν που είχε το Κοινοβούλιο. Τώρα, πια, δεν θα χρησιμοποιούμε δογματικά το μακροπρόθεσμα. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα βήματα για να υιοθετήσουμε ένα καθεστώς χωρίς θεώρηση. Ξέρω ότι είναι περίπλοκο το θέμα και ξέρετε κι εσείς ότι η αντιπροσωπεία μας έχει ετοιμάσει ένα λεπτομερές έγγραφο μέσα στο οποίο αναλύουμε με ποιο τρόπο λειτουργεί σήμερα το καθεστώς των θεωρήσεων. Έχουμε μιλήσει για τις αρνητικές συνέπειες που έχει το καθεστώς αυτό στην ε, μετακίνηση ανθρώπων και στις επαφές της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο έγγραφο αυτό καταδεικνύουμε ότι είναι λιγότεροι οι Ουκρανοί σήμερα που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι κατά το παρελθόν. Είναι οι θεωρήσει, το σύστημα αυτό, το οποίο αποτελεί ένα φραγμό, ένα εμπόδιο στον να έρχονται Ουκρανοί στην Ευρώπη. Είναι και πολιτικό εμπόδιο. Πιστεύω λοιπόν ότι οι θεωρήσεις έχουν σαν αποτέλεσμα να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Ουκρανοί, ακόμα και να σχηματίζουν αρνητική γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν οι εκλογείς οι Ουκρανοί ε, πάνε στις κάλπες και αποφασίζουν ε, για το ποιος θα τους εκπροσωπήσει, ψηφίζουν έχοντας την ε, εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υπέρ της Ουκρανίας. Όσο σιωπούμε για το θέμα αυτό των θεωρήσεων, ή όταν είμαστε δογματικοί για το ζήτημα αυτό, αυτό έχει αρνητικές συνέπειες. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που η προσέγγιση αυτή αλλάζει και το είδα. Το είδα μάλιστα όταν ο Επίτροπος πήρε το λόγο στην τελευταία συνάντηση που είχαμε, η αντιπροσωπεία μας δηλαδή, και το είδα και στον τρόπο που ε, μας μιλήσατε εσείς σήμερα για το καθεστώς χωρίς θεωρήσεις. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε ακόμα με την Ουκρανική πλευρά για να καταλήξουμε κάπου υπέρ ενός καθεστώτος χωρίς θεωρήσεις. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω να μου ξεκαθαρίσετε ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ώστε να μπορέσουμε τελικά να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σύστημα καθεστώτος χωρίς θεωρήσεις. Ίσως θα έπρεπε να προβλέψουμε την εκπόνηση κάποιου γράφου για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι λέτε. Το θέμα των θεωρήσεων, επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και θα μας βοηθήσει η κατάργηση στις στενότερες σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Όσον αφορά τώρα τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, εδώ θα ήθελα να ξέρω ποιες θα είναι οι συνέπειες από την εισαγωγή στην Ουκρανία πολύ συγκεκριμένων διατάξεων για τις μεταφορές, για τα τελωνία και για τη γεωργία ιδιαίτερα. Εγώ αναρωτιέμαι και δεν την έχω την απάντηση, γι' αυτό και σας ρωτάμε εσάς. Δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να βρούμε πολύ συγκεκριμένα τι επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά πάνω στους Ουκρανούς παραγωγούς. Γιατί εμεί κάνουμε διαπραγματεύσεις για διάφορες διατάξεις, χωρίς όμως να γνωρίζουμε καλά ποιες θα είναι οι συνέπειες στην Ουκρανία από αυτές. Επίσης πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουν υπόψη τους οι Ουκρανοί παραγωγοί τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν πρέπει να εφαρμόσουν νέους κανόνες, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχουν καμία προοπτική μακροπρόθεσμα, αυτό θα είναι δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Διευθυντά, θέλω να σα ρωτήσω, υπάρχουν αναλύσεις, υπάρχουν ε, μελέτες που έχουν γίνει για τις συνέπειες, τις οικονομικές, για παράδειγμα, που θα έχει εφαρμογή των κεφαλαίων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στην Ουκρανία, στους Ουκρανούς. Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε. Υπάρχουν ενδεχομένω απειλές για το μέλλον από μια τέτοια κατάσταση. Κάτι άλλο στο οποίο θέλω να αναφερθώ τώρα. Πραγματικά, δεν ξέρω την ημερομηνία πότε θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει. Η αλήθεια είναι ότι δίστανται οι απόψει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μερικέ φορέ μα λέει ότι προχωρούν διαπραγματεύσει γοργά, ότι υπάρχει βούληση από πλευρά τη Ουκρανία, αλλά εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθούν. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να δώσει κάποιο μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να ξέρουμε λίγο πολύ. Θυμάμαι ότι επί Σουηδική προεδρία μας είχαν πει 6 μήνες. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπήρξαν εκλογέ στο μεταξύ εκεί και γι' αυτό καθυστέρησαν τα πράγματα, αλλά σήμερα μιλάμε για 12 μήνες. Φυσικά και πρέπει κάποιες προϋποθέσεις να υπάρχουν για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Όμως γι' αυτό θέλω να ξέρω. Ποιο είναι ο λόγος για τον οποίο η ημερομηνία κατάληξης των διαπραγματεύσεων απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Γιατί, ενώ η κατάσταση είναι αρκετά θετική, όλα αυτά η ημερομηνία κατάληξης αναβάλλεται συνεχώς. Τέλος, κάτι άλλο που με ενδιαφέρει όλος και θέλω να γνωρίζω εσείς πώς εκτιμάτε την κατάσταση όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική της Ουκρανίας. Ορισμένα θεσμικά όργανα που ασχολιόντουσαν στην Ουκρανία με την πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αλλάξει ή ακόμα και έχουν καταργηθεί. Νομίζω ότι υπάρχει μια επιτροπή που καταργήθηκε στην Ουκρανία. Από την άλλη μεριά όμως μας έρχονται πολύ θετικά μηνύματα από την Ουκρανία τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό και εγώ δυσκολεύομαι να ερμηνεύσω την, τον προσανατολισμό της Ουκρανίας σήμερα. Ποιο είναι αυτός ο προσανατολισμός της Ουκρανίας λοιπόν σήμερα και ειλικρινά ποια είναι η δικιά σας συγγνώμη βάσει τη δικιάς σας εμπειρία στο θέμα. Κατά τη γνώμη σας, προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουν οι αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της Ουκρανίας και ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική της Ουκρανίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν περάσει ήδη αρκετές εβδομάδες μετά τις εκλογές και τον νέο πρόεδρο. Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποια πρώτα συμπεράσματα, έτσι δεν είναι, ακόμα και αν αυτό είναι λίγο δύσκολο. Θέλω λοιπόν παρακαλώ να μου πείτε ποια είναι η δικιά σας γνώμη για το θέμα. Συνοψίζω. Θεωρήσεις, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Στη συνέχεια, συνέπειες της εφαρμογής των κανόνων που περιλαμβάνονται στην συμφωνία και κατάληξη, ημερομηνία καταληκτική για τις διαπραγματεύσει. όπως επίσης τέλος οι αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της Ουκρανίας, ιδιαίτερα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιε είναι. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Πρόεδρος, πρέπει τώρα να δώσω την προεδρία στον κύριο Πασκού και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Ε, θα επανέλθω αύριο το πρωί. Γεια σας. Κύριε Μιγκαρέλ, θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Κοβάλη για αυτές τις 4-5 ερωτήσεις. Μπορώ να σας απαντήσω σε μία μόνο πρόταση, πολύ εύκολα. Η πρώτη ερώτησή σας ήταν για την μετακίνηση των ατόμων. Θα συνοψίσω ως εξής την τωρινή κατάσταση. Η Ουκρανία εδώ και τρία χρόνια υλοποιεί μια συμφωνία για την διευκόλυνση για την έκδοση θεωρήσεων για τις βραχυπρόθεσμες διαμονές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μια συμφωνία για την επανεισδοχή των παρανόμων διαμενόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν συλληφθεί. Παράλληλα με την υλοποίηση αυτών των δύο συμφωνιών που διευκολύνουν λοιπόν την έλευση στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιων κατηγοριών ε, ε, Ουκρανών υπηκόων, οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δρομολόγησαν σε συνεργασία με τους ομολόγους μας μια συμφωνία για τη θεώρηση, ούτως ώστε να προσδιορίσουμε τους όρους που θα μας επιτρέψουν εν ευθέτω χρόνο να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις και να οδεύσουμε προς την απελευθέρωση για τις θεωρήσεις. Ποιες, ποιοι είναι οι όροι για να ε, επιτύχουμε την ελεύθερη κυκλοφορία. Οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπαμε, συζητούν με τους ε, Ουκρανούς ομολόγους τους για τους όρους με τους οποίους πρέπει να συμμορφωθεί η Ουκρανία, ούτω ώστε να προωθήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία. Και σχετίζονται αυτοί οι όροι με τα εξή στοιχεία. Πρώτον, διαχείριση των συνόρων. Δεύτερον, ε, την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων. Τρίτον, την πολιτική ε, μετανάστευση σε θεωρήσεων και ασύλου. Τι επιθυμούν σήμερα οι Ουκρανοί να αποκτήσουν ένα οδικό χάρτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως παραδείγματος χάρη αυτός που είχαμε με κάποιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και που οδήγησαν ε, σπευσμένα στην ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό λοιπόν θέλουν και οι Ουκρανοί. Και τώρα συζητείτε το θέμα στο Συμβούλιο ε, για να δούμε αν αιτιολογείται η χορήγηση τέτοιου οδικού χάρτη στην Ουκρανία για να επιτύχουμε την ελεύθερη κυκλοφορία. Και θα τα ξαναπώ για να είμαι σίγουρο θα με καταλάβετε. Οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται ε, με τους Ουκρανούς για τους όρους που, με τους οποίους πρέπει να συμμορφωθεί η Ουκρανία για να επιτύχουμε την ελεύθερη κυκλοφορία. Ταυτόχρονα γίνεται συζήτηση στο Συμβούλιο σχετικά με τη δυνατότητα χορήγηση στην Ουκρανία ενό οδικού χάρτη που θα οδηγήσει στην ελεύθερη κυκλοφορία. Καταλαβαίνετε, διακυβάβεται. Αν υπάρξει οδικός χάρτη, υπάρχει αυτοματοποίηση τη διαδικασία. Με το που πληρούνται οι όροι, εφαρμόζεται ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό έγινε σχάντω με τρει χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Αν δεν υπάρχει οδικό χάρτη, αν υπάρχει μόνο διάλογο για τι θεωρίε όπω αυτό που γίνεται τώρα,

Ε, υπάρχει αυτό το στοιχείο της πολιτικής κρίσης ε, για να διαπιστώσουμε το εξή Με το που υπάρξει συμμόρφωση με τους όρους, ενδείκνεται ναι ή όχι να προχωρήσουμε στην ελεύθερη, στην ελεύθερη κυκλοφορία. Δεύτερον, για τη ζώνη ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών. Ναι, πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων έγινε αξιολόγηση αντικτύπου για, τις για τους διαφόρους τομείς της οικονομίας της Ουκρανίας σχετικά με την εγκαθίδρυση ζώνης, ε, πλήρους ζώνης ζώνης ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών που αποτελείται από δύο στοιχεία. Πρώτον, να καταργήσουμε ό,τι υπολείπεται από τους τελωνιακούς εφραγμούς. Η Ουκρανία ξέρετε ότι ανήκει ε, στον ΠΟΕ και δύο χρόνια, άρα δεν υπάρχουν πολλοί φραγμοί και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης ε, συζητήθηκε και το θέμα της κατάργησης ε, των τελωνιακών φραγμών. Ε, υπάρχουν όμως οι μη δασμολογικοί φραγμοί, δηλαδή η ε, ρυθμιστική σύγκληση, η κανονιστική σύγκληση. Να μεριμνήσουμε λοιπόν ώστε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζονται από την Ουκρανία. Αυτό φυσικά χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Δεν είμαι σε θέση τώρα ε, να σας πω πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι Ουκρανοί για να ενστερνιστούν να εφαρμόσουν τα πρότυπα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό εξαρτάται από τη συνέπειά, από τη σχολαστικότητά τους και από τους διοικητικούς τους περιορισμούς. Τώρα, ω προ τον αντίκτυπο για την οικονομία της Ουκρανίας ε, δεν δυνάμεθα να κάνουμε συνολική αξιολόγηση. Τι συμβαίνει. Ε, σε ένα πρώτο στάδιο υπάρχει, υπάρχουν προσαρμογές όπου πλήττονται διάφοροι οικονομικοί τομείς. Ε, ποιοι είναι αυτοί οι τομείς, δεν είναι τομείς. Άνθρωποι πλήττονται που εργάζονται μέσα σε επιχειρήσεις ε, που ε, τύχαν προστασίας από τον διεθνή ανταγωνισμό και συγκεκριμένα τον διεθνή ανταγωνισμό των δικών μας εμπορικών φορέων πλέον δεν προστατεύονται, γίνονται αυτές οι προσαρμογές επώδυνες και βραχυπρόθεσμα θα πληγεί η οικονομία ε, της Ουκρανίας μέσω μακροπρόθεσμα. Αν αυτό συνδυαστεί με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εμείς προκρίνουμε, είναι σαφές ότι η ουκρανική οικονομία θα βγει κερδισμένη τελικά. Ε, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναβαθμιστεί το επίπεδο διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Οπότε ε, δίνω ασαφή απάντηση γιατί δεν είμαι σε θέση να σας δώσω σαφέστερη απάντηση. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω τελικά ποιοι τομείς θα υποφεληθούν από το άνοιγμα των αγορών και πότε. Ε, στην αρχή η βραχυπρόθεσμα σας λέω είναι πόδινη η προσαρμογή και μέσω μακροπρόθεσμα είναι ευνοϊκή. Τώρα, για την ημερομηνία περάτωσης, ε, ε, Α πάρουμε τα πολιτικά κεφάλαια, τα κεφάλαια τομιακής συνεργασίας και τα κεφάλαια που άπτονται τη ελευθερία ασφάλεια και δικαιοσύνη, όπω λέμε εμεί, Ε, λοιπόν μα χρειάζονται δύο-τρει εβδομάδε. Ε, ε, στο πολιτικό τομέα τι γίνεται. Έχουμε την προοπτική προσχώρηση, αυτό είναι σαφές, δεν χρειάζεται. Σε ένα λεπτό μπορούμε να του δώσουμε την απάντηση. Για την ελεύθερη κυκλοφορία ε, είναι λίγο πιο ασαφή τα πράγματα, αλλά δεν θα χρειαστούμε πολύ χρόνο στην Ένωση για να αποφασίσουμε τελικά ε, οι μακροπρόθεσμες ή όχι προοπτικές και για την ελεύθερη κυκλοφορία ισχύουν. Και τέλο, υπάρχει το θέμα τη εδαφική ε, ακαιρεότητα. Πρέπει να κατανοήσει η Ουκρανία ότι δεν είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατοχυρώσει την ασφάλεια οποιοδήποτε εξωτερικού εταίρου. Εντάξει, μπορούμε να μεριμνήσουμε ε, ούτως ώστε οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στα πλαίσια διεθνών οργανισμών τελικά θα τηρηθούν για την εδαφική κυριαρχία, για την εδαφική ακεραιότητα αλλά ε, ποια έχει να, να δώσουμε για την ασφάλεια. Ε, για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη λοιπόν χρειαζόμαστε δύο-τρει εβδομάδε. Το βασικό πρόβλημα είναι το εμπορικό κομμάτι και είναι βασικό το πρόβλημα γιατί είναι πολύ πιο τεχνικές οι διαπραγματεύσεις. Σας είπα από τα 14 κεφάλαια, τρία έχουμε κλείσει προσωρινά, υπολείπονται άρα 11 και μου λέτε ότι οι Προεδρία σε ανακοίνωσαν τη λήξη για το επόμενο εξάμεινο και τώρα σας λέω θα πάρει από 6 έως 12 μήνες. Ναι, αλλά στην προεκλογική του εκστρατεία ανέλαβαν περιοριστικά μέτρα για τι εμπορικέ συναλλαγές και μέτρα που αντιβαίνουν στις δεσμές που έχουν λάβει στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Οπότε αυτό περιπλέκει ε, τις ε, διαπραγματεύσεις που θα κάνουν μαζί μας για τις ε, συμφωνίε ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών. Από αυτού, εξαρτάται. Αν δείξουν αποφασιστικότητα αύριο, αν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, από 6 έως 12 μήνες, να, αυτή η περίοδος νομίζουμε θα χρειαστεί, αλλά πιο σαφής δεν μπορώ να κάνω, γιατί αλλιώς θα αρχίσω ε, να τεκμέρω πράγματα και δεν νομίζω να σα βοηθάει αυτό. Ε, τώρα, από τι έγινε από τις τελευταίες εκλογές και ποια, ποιο είναι το αποτελέσμα της αξιολόγησης που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, λοιπόν, ο Πρόεδρος είπε αυτά που περιμέναμε. Επανέλαβε ότι κατά τη γνώμη του ο προευρωπαϊκός ε, προσανατολισμός της χώρας του παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για αυτόν. Επιβεβαίωσε Ε, ότι ο Πρωθυπουργό Τίμκο, που γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί εδώ και 15 χρόνια ε, ήταν υπουργό παρά το Πρωθυπουργό και ασχολείται με την οικονομία και τι σχέσει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και ο Κωνσταντίν Ρισέσκο, υπουργό εξωτερικών, που επίση γνωρίζουμε πολύ καλά και που ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει η χώρα για να οδεύσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ε, με αυτούς τους διορισμούς, έτσι να πω, καλά είναι τα νέα. Ε, και πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τις δηλώσεις του κυρίου Κόβιτσε. Αλλά δεν θα ήμουν απολύτω ειλικρινή αν σας έλεγα ότι δεν υπάρχουν και κάποια κάπως ανησυχητικά στοιχεία. Να αναφέρω δύο μόνο. Ξέρετε ότι ασκείται κάποια πίεση στην Ουκρανία ούτω ώστε να προσχωρήσει στην Τελωνιακή Ένωση αυτή η χώρα της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν δηλαδή. Εάν ε, καρποφορήσει η πίεση, αν προσχωρήσει αυτή την τελωνιακή ένωση η Ουκρανία, ε, τότε δύσκολα θα μπορέσει να δημιουργήσει η τελωνιακή ένωση η Ουκρανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αν προσχωρήσει την άλλη τελωνιακή ένωση, τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Θα έχει κοινό εξωτερικό δασμό η Ουκρανία με τρεις χώρες, ε, των οποίων οι συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν απελευθερωθεί παρά μόνο λίγο. Οπότε θα βρεθούμε σε μία στενοπό και το ξέρουν. Ξέρουν ποιες θα είναι οι συνέπειες της προσχώρησής τους σε αυτή την τελωνιακή ένωση. Από την άλλη είμαστε σαφείς στις σχέσεις μας όταν συζητούμε αυτό το θέμα με την Ουκρανία. Τι σημαίνει μια τέτοια προσχώρηση. Δεύτερο ανησυχητικό στοιχείο. Τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο. Ξέρουμε ότι διαπραγματεύονται οι Ουκρανοί με τους Ρώσους ε, για την αναθεώρηση της συμφωνίας ε, σχετικά με την αγορά ε, του ελεύθερου αερίου από την Ουκρανία που βάσει της συμφωνίας που την Τιμοσέκο της, του 2009. Ξέρουμε επίσης ότι οι Ρώσοι έχουν θέσει κάποιους όρους για να αρχίσει να ισχύει και πάλι αυτό το συμβόλαιο. Ποιοι είναι αυτοί, μεταξύ άλλων δημιουργία ενδεχομένως μιας κοινοπραξίας. Ε, και φυσικά δεν θα είναι μακριά από την με αυτή την κοινοπραξία και ε, θα έχει το λόγο της ε, στη διαχείριση του δικτύου, τόσο ώστε να περνάει το ρωσικό αέριο από την Ουκρανία για να φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί θα μπορούσαμε, μπορεί να ανακύψουν προβλήματα. Λοιπόν, συνοψίζω, ε, είναι καθησυχαστικές οι δηλώσεις, ε, υποστηρίζονται από το διορισμό ικανών ανθρώπων ε, που είναι αποφασισμένοι να οδεύσουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν βρίσκεται σε ένα πολιτικό κενό η Ουκρανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που την πιέζουν, οι οποίες δεν την πιέζουν απαραίτητα προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά μπορώ να σας απαντήσω προς το παρόν. Τώρα λοιπόν ε, θα ξεκινάει ένας ε, διμερής διάλογος. Ε, μία ερωτησούλα μόνο. Ε, εάν τελικά εγκριθεί ο δικός χάρτης, έχουν προβλεφθεί όροι για την έγκριση αυτή του οδικού χάρτη. Υπάρχουν προϋποθέσεις για την έγκριση του οδικού χάρτη. Γνωρίζετε κάτι παραπάνω γι' αυτό ή ε, πρόκειται ε, για δύο παράλληλες διαδικασίες, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν στην Επιτροπή και η συζήτηση στο Συμβούλιο. Ε, και ποια, ποιες είναι οι πιθανότητες έγκριση οδικού χάρτη. Απάντηση. Όχι, προϋποέθεση δεν υπάρχει. Είναι πολιτική συζήτηση προς το παρόν. Το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει ε, αν ενδείκνυται να χορηγεί στην Ουκρανία, όπως έκανε πριν από λίγους μήνες σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τον οδικό αυτό χάρτη ή όχι. Μα πολιτική απόφαση είναι. Ε, το Συμβούλιο θα αποφασίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δική της άποψη προφανώς, αλλά αποφασίζει το Συμβούλιο. Well, thank you. Mr. Severin, please. Well... Κύριο Σεβερέν. Μετά από αυτή την ε, μακρά εισαγωγή, κατ' ουσίαν δεν υπάρχουν ε, ερωτήσεις, απλά θα ήθελα να έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων. Βλέπω λοιπόν ότι προκύπτουν πολλές ευκαιρίες στη σχέση μας με την Ουκρανία δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία και αυτό όχι διότι υπήρξαν ε, ουσιαστικές αλλαγές στην Ουκρανία, αλλά κυρίως διότι αυτή η κατά τα άλλα η συνήθως ε, φυσιολογική εναλλαγή στην εξουσία, κάτι που είναι αρκετά απλό και φυσιολογικό στις ε, δικές μας τις χώρες, μας ε, θυμίζει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτές τις ε, δογματικές και μανιχαϊστικές απόψεις που είχαμε κατά το παρελθόν και τώρα ε, θα πρέπει να υπάρχει μια φιλοουκρανική κυβέρνηση, οχι φιλορωσική ούτε φιλοευρωπαϊκή. Διότι όσο η ηγεσία αυτή φιλοουκρανική, κατά την άποψή μου θα αναζητήσει ελευθερία και ανάπτυξη στη χώρα. Και όποιος ψάχνει να βρει κάτι τέτοιο, κατά άποψή μου, είναι φιλοευρωπαίος. Ε, βεβαίως και πρώτα απ' όλα είναι προφιλοουκρανός. Αυτό όμως ε, απαιτεί ε, από την πλευρά μας να είμαστε και πιο τολμηροί. Και πρέπει τρεις βασικές απόψεις να τις προάγουμε, μεταξύ αυτών την πολιτική σύγκληση. Παράλληλα, Θεωρώ ότι πρέπει να ε, προχωρήσουμε με την ε, πολιτική δύο κατευθύνσεων, να έχουμε διμερείς ε, συζητήσεις για την ζώνη ελεύθερων ανταλλαγών, γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν δύο ζώνες ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών. Και για να τελειώσω θα ήθελα να πω ότι πράγματι πρέπει να περάσουν τρία σαφή μηνύματα. Το ένα είναι πρακτικό, ότι θα πρέπει να διτεθεί το δεύτερο πακέτο ε, βοήθειας προς την Ουκρανία, γιατί αν δεν βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, τότε κατά την άποψή μου αυτό θα είναι ε, το πρώτο βήμα στο να χάνουμε την ευκαιρία. Δεύτερον, όσον αφορά τον χάρτη πορείας, ε, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να περάσουμε ένα ευκρινές μήνυμα στο Συμβούλιο και ας είμαστε ειλικρινεί, υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία διαφωνούν και αυτά δημιουργούν προβλήματα. Αυτός λοιπόν ο χάρτης πορεία καθαρά τεχνικά, όπως το ανέφερε και η δική μα η αντιπροσωπεία, μπορεί η βίζα, η θεώρηση, αναφέρομαι στο νέο καθεστώς θεωρήσεων, μπορεί να προσφερθεί, να τους δοθεί ε, μετά από λίγα χρόνια, όχι τόσο μακροπρόθεσμα. Τέλος, ε, νομίζω ότι θα πρέπει ε, να ξεφύγουμε από το αμφιλεγόμενο των ε, προοπτικών. Να είναι σαφείς οι προοπτικές. Είναι μια χώρα επιλέξιμη για υποψηφιότητα και θα μπορούσαν να γίνουν μέλη αν επιτύχουν πράγματα. Ενεργειακή Ένωση, Ζώνη Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών, καθεστώς απελευθέρωσης των ε, θεωρήσεων, όλα αυτά πριν de καταστούν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, αναφέρθηκε μία προσπάθεια να καταδειχθεί ο χάρτης προς την κατεύθυνση της ένταξης. Και εμείς ε, Είπαμε ότι θα μπορεί να είναι κατεύθυνση ε, προς την ένταξη, μπορεί και προς κάτι άλλο. Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι κρύβεται πίσω από μια διπλωματική γλώσσα. Ε, υπάρχουν ε, κάποιες επιτυχίες και οι Ουκρανοί έχουν επιδείξει κάποιο αίσθημα ευθύνης. Πάντως πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε πλέον μία ομάδα η οποία μπορεί να εφαρμόσει μια συνεπή πολιτική. Έχουμε τον πρόεδρο, έχουμε ε, κοινοβουλευτική πλειοψηφία και έχουμε και συνομιλητή. Κάποιον που μπορεί να δεχθεί τις ερωτήσεις ε, για τις κοινοτικές πολιτικές. Και δεν είναι μόνο έτσι αέρας και λόγια από πλευράς Ουκρανίας. Τώρα πλέον ε, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο όπου μπορούμε να προχωρήσουμε. Και έχει φτάσει πια η χρονική στιγμή έτσι ώστε και εμείς ε, να είμαστε ειλικρινείς σε αυτά που λέμε. Να ξεφύγουμε από αυτήν την αντιευρωπαϊκή ε, μεγαλοστομία που υπήρχε αυτό βιώσαμε τα τελευταία χρόνια. Ο πρόεδρος Γιαννόκοβιτς σε μια σύντηση που είχα μαζί του πριν από μια εβδομάδα είπε με απόλυτη σαφήνεια ότι φοβούνται ότι οι άνθρωποι ε, μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς οι Ουκρανοί να γνωρίζουν ποιες θα είναι οι πρακτικές επιπτώσεις στους ίδιους. Και είπε ότι δεν, ξέρει, δεν ξέρουν ακριβώς ε, τι πρέπει να κάνουν. Για το θέμα των θεωρήσεων αυτό είναι πολιτικής φύσης θέμα, δεν είναι απλά διοικητικό ή τεχνικό. Διότι για να υπάρξει πρόοδος στις ε, θεωρήσεις, μάλλον αν υπάρξει πρόοδος, αυτό θα έχει σημαντική ε, επίπτωση στην κοινωνία της Ουκρανίας. Όπως γνωρίζει και την προσωπή και ο κύριος Κόβα, τώρα πλέον έχουμε φτάσει σε μια τέτοια, φάση όπου οι αιτήσει ε, για θεωρήσεις ε, είναι μόνο σε ένα 4%. Δεν είναι απλά στατιστικό ποσοστό, έχει και πρακτικές συνέπειες το μόνο το 4% των αιτήσεων αφορούν τη χορήγηση βίζα θεώρησης. Ο κύριος Λαμπερίς. Νομίζω ότι όλοι εδώ καταλαβαίνουν και συμφωνούν ότι η νέα ηγεσία της Ουκρανίας δεν έχει τρίτη επιλογή ή που θα μπει στην Τελωνιακή Ένωση της Ρωσίας ή που θα αφήσει ανοιχτή την πόρτα προς μια ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την ε, Ευρώπη. Η Ουκρανία δεν λέει όμως. Θα συνεχίσει να θέλει δεσμούς με την Ευρώπη. Οπότε τότε δεν θα μπει στην Τελωνική Ένωση με τη Ρωσία γνωρίζουν πλήρως, ξέρουν, είναι προειδοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημερωμένοι για το ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέραν από αυτές τις δύο. Είναι εν γνώση. Ο κύριος Κοβάτσεφ τώρα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον ε, δοκτόρα Μιγκαρέλη, τον κύριο Μιγκαρέλη για τόσα μας είπε. Εγώ εκ μέρους του ΕΛΚ θέλω να πω ότι το ΕΛΚ στηρίζει απόλυτα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ουκρανίας. Έχουμε κοινή ιστορία με αυτή τη χώρα, κοινέ αξίες και χαιρόμαστε για τις εκλογές που έλαβαν χώρα πρόσφατα και που κρίθηκαν από τους παρατηρητές τόσο τους διεθνείς όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίκες και σωστές. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Πρώτον, σε αυτό το πρώιμο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η νέα κυβέρνηση, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν ε, αλλαγές όσον αφορά την τακτική που ακολουθεί η νέα κυβέρνηση στις διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, θα ήθελα να ήξερα Ποια από τις προτεραιότητες που υπάρχουν για το 2010 πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει περισσότερες ε, δυσκολίες στο θέμα του δικαστικού συστήματος, η, η εφαρμογή του εθνικού σχεδίου κατά της διαφθοράς. Ξέρουμε ότι οι προβλήματα υπάρχουν και εδώ στον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς αξιολογεί τη συμμετοχή της Ουκρανίας ε, στη συμφωνία για την ενέργεια. Ξέρετε ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο κάποιος ανταγωνισμός. Δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για την εταιρική σχέση, οπότε μπορούμε να πούμε ότι η Ουκρανία προσανατολίζεται περισσότερο στην ανατολική εταιρική σχέση. Προσθέθηκε και ο κύριος Τάνοκλη, ο πρόεδρος, τελευταίος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Γρήγορα, ερώτηση προς την Επιτροπή. Ε, μίλησα με έναν δημοσιογράφο, πήρε τηλέφωνο, ένας δημοσιογράφος από το Κίεβο, που ήθελε να σχολιάσω ε, την άποψη της Κομισιόν. Και εγώ είπα, ας πάρω καλύτερα τηλέφωνο την Γενική διεύθυνση Ενέργειας. Βλέπετε στο Κίεβο κυκλοφορεί ιστορία για την κυβέρνηση, ε, ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ενέργειας ότι ετοιμάζονται για συμφωνία με τον κύριο Φέρτας που ήταν ε, ο κύριος μέτοχος στο Ρώσο-Ουκρανέγκο αυτή την ιστορία ε, για την οποία φρόντισε να διαλύσει αυτό το όργανο προηγούμενη κυβέρνηση που στήχησε εκατομμύρια για να πω δισεκατομμύρια δολάρια είχε να κάνει με τη ρωσική Κασπρόμ και τους Ουκρανούς καταναλωτές και τώρα από ό,τι κυκλοφορεί στο Κίεβο η νέα κυβέρνηση θέλει τον κύριο Φέρτης που χρηματοδότησε την εκστρατεία του Πρόεδρου Γιαννέσκου να το επιτρέψει λοιπόν η νέα κυβέρνηση να αγοράσει ένα μεγάλο ποσοστό του Ουκρανικού συστήματος αγωγών είτε αγοράζοντας νέους αγωγούς είτε ή φτιάχνοντας νέους αγωγούς ή αγοράζοντας άλλους που ήδη ανήκουν στο Ουκρανικό κράτος. Κυκλοφορεί επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Κομισιόν έχει αντιτεθεί στην ιδέα αυτή. Γιατί σημαίνει ότι εκεί εμπλέκονται και κοινοτικά χρήματα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Εσείς μπορείτε να σχολιάσετε ή δεν έχετε ιδέα. Και αν έχετε ιδέα, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κοιτάζει. Ευχαριστούμε. Τώρα μπορείτε να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ. Έφυγε εμένα ο κύριος Σεβερίν, αλλά εγώ θα απαντήσω στην ερώτηση του. Λέει ότι δεν χρειάζεται αντιπαράθεση με τις νέες αρχές. Εννοείται. Είναι προφανές. Ο πρόεδρος Γιαννουκοβίτς εξάλλου ξέρουμε ότι έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία δέκα χρόνια. Έχει αλλάξει. Και ότι η δεύτερη φορά που ήταν ε, ε, ο Πρωθυπουργό ήταν ε, εντελώ διαφορετικό από ό,τι όταν ήταν την πρώτη φορά Πρωθυπουργό. Τη δεύτερη φορά ήταν πολύ διαφορετικό. Η υποκυβέρνηση Γιαννούκοβιτ 2, μην ξεχνάμε, η Ουκρανία πέρασε 21 νόμους που την βοήθησαν να μπει στον ΠΟΕ. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να υποψιαζόμαστε τις νέες αρχές της Ουκρανίας, καθ' άλλο. Όπως είπατε, Άνθρωποι όπως ο πρόεδρος Γιαννούκοβιτς ή ο πρωθυπουργός Λαζαρόφ, ο υπουργό εξωτερικών Ιεσέγκο, είναι άνθρωποι ε, οι οποίοι φέρνουν αποτελέσματα, κάνουν, τηρούν το λόγο τους και κάνουν ό,τι υποσχέθηκαν. Οπότε έχουν πει ότι θέλουν προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου, είδαμε τη, τα αποτελέσματα των εκλογών σαν μια ευκαιρία για μας να ενισχύσουμε την προσέγγιση με αυτή τη χώρα. Για τα τρία ξεκάθαρα μηνύματα που θέλει ο κύριος Σεβερή να περάσουμε. Αρρωγή, πρώτα απ' όλα, για να βγουν από την οικονομική κρίση. Έχουμε ετοιμάσει μία μακροοικονομική με βοήθεια με 600 εκατομμύρια που θα αποδεσμευτεί, εφόσον συμφωνήσετε, μόλις η Ουκρανία θα προσαρμοστεί με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή μήνες. Η ελεύθερη διακίνηση. Μίλησα για αυτή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο. Και για τις προπτικές ένταξης προς το παρόν είναι ένα ζήτημα που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Το άρθρο πάντως 49 της συνθήκης λέει ξεκάθαρα ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για κάθε ευρωπαϊκή χώρα η οποία τηρεί κάποιες προϋποθέσεις, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός των μειονοτήτων, για παράδειγμα. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο η Ουκρανία, οπότε έχουν πέρασει τρία χρόνια διαπραγματεύσεων. Δεν μπορούν να κρυθούν επιτυχή. Ε, τι να πω, θα μπορούσαν να ήταν και καλύτερα. Όπως σας είπα, ήδη τον πρώτο καιρό προχωρήσαμε με το πρόγραμμα δράσης για την καλλιγυθνίαση. Μετά σε λίγους μήνες ετοιμάσαμε την ατζέντα για την σύνδεση. Ήδη αυτά τα δύο έγγραφα πήραν πολύ χρόνο και αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Ε, από εκεί και πέρα είναι μια συμφωνία η οποία σύμφωνα με τους ειδικού για τα νομικά και θεσμικά ζητήματα που είναι από τις πιο περίπλοκες που έχουν διαπραγματευτεί μέχρι τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα χρειάζεται και χρόνος. Έρχομαι τώρα στην ερώτηση του κύριου Λανμπέργκης. Κατά πόσο ξέρουν τι θα σήμαινε για αυτούς το να μπουν σε τελωνιακή ένωση με τους γείτονές τους στη Ρωσία. Ναι, το ξέρουν. Τους το έχουμε εξηγήσει με λεπτομέρειες, οπότε ξέρουν πολύ καλά. Και τελευταία ερώτηση ήταν για την μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα και τα μέτρα κατά της διαφθοράς. Έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά σε αυτούς τους δύο τομείς τα τελευταία χρόνια, αλλά μένουν και πολλά ακόμα να γίνουν. Είναι δύο μεταρρυθμίσεις που πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την Ουκρανία τους επόμενους μήνες. Ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δικαστών και βέβαια και διπλασιασμός προσπάθειων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Εξάλλου δεν είναι η μόνη χώρα που πρέπει να κάνει προσπάθειες σε αυτούς τους τομείς. Τώρα η εμπλοκή της Ουκρανίας ε, για την Μαύρη Θάλασσα. Ε, η Ουκρανία και το Κίεβο. Θα δουν εμείς να πούμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν πόροι ακόμα και αν είναι περιορισμένοι. Τώρα αν υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στην συνεργεία Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Εταιρική Σχέση ε, δεν υπάρχει η συνεργία Μαύρη Θάλασσα είναι περιφερειακή συνεργασία γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα για τους συγκεκριμένους τομείς που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά, την ενέργεια και το περιβάλλον και η ανατολική εταιρική σχέση είναι πώς οι έξι εταίροι μας θα προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς. Πρόκειται λοιπόν για δύο πρωτοβουλίες οι οποίες δεν επικαλύπτονται. Και γι' αυτό πρότεισε ο κύριος Στάνοκ. Ναι, γνωρίζουμε ότι οι ιδιοκτήτες που η Γιούλια Τιμοσέγκο τους ε, πήρε ζητούν αποζημίωση για ένα μέρος των αποθεμάτων φυσικού αερίου που από ό,τι είπαν τους ε, τα πήρε η προηγούμενη κυβέρνηση και θέλουν αποζημίωση. Ξέρετε και γνωρίζετε πολύ καλά την Ουκρανία, όπως και εγώ, ότι ορισμένοι πρόσωποι από τους πρώην ιδιοκτήτες σήμερα κατέχουν υπεύθυνε θέσεις. Γιατί ακριβώς όπως το είπατε, οι απαλλατρώσεις αυτές έγιναν ε, σε ορισμένους οι οποίοι χρηματοδότησαν την προκλογική εκστρατεία του σημερινού Πρόεδρου μπορείτε να είσαστε βέβαιος ότι χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα πάνε για τη χρηματοδότηση της φυρτάς. Αυτό είναι βέβαιο. Και δεύτερον, έχουμε περάσει ξεκάθαρα μηνύματα προς τις Ουκρανικές αρχές και τον Υπουργό Μποϊκό, ώστε να μην ληφθούν παράλογα μέτρα σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστώ εσάς και όλους τους υπόλοιπους και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η κατάσταση στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στις 3 Οκτωβρίου Είχαμε εκλογές, ε, έχουμε πολιτικό αδιέξοδο και εξακολουθούν να, εξακολουθούμε να περιμένουμε την ε, τοποθέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Κυρία Πακ, κοιτάξτε, πριν από ένα χρόνο κατέθεσα μία έκθεση και θα μπορούσα να πάρω αυτή την ίδια έκθεση ίσως λίγο πολύ, αλλά εν τω μεταξύ τα πράγματα επιδεινώθηκαν πλέον δεν είμαστε σε κατάσταση όπου να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι βελτιώθηκε το πολιτικό καθεστώς, ότι οι πολιτικοί συνετίστηκαν. Κάθε άλλο είμαστε αναγκασμένοι να συνειδητοποιήσουμε την έλλειψη βούλησης. Η ε, κατάσταση που στην Ερσεγοβίνη δεν μοιάζει να βελτιώνεται στο μέλλον. Προκύπτει λοιπόν πολιτική ε, αποτελμάτωση και βλέπουμε ότι ε, εκφράζονται όλο και μεγαλύτερες ε, εθνικιστικές κορώνες και όχι μόνο διότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Οι κορώνες αυτές εκτοξεύθηκαν και πέρυσι και πρόπερσι και εκφράστηκαν μάλιστα και αρκετά οξύες απειλές από τη Ρεπούμπλικα Σπέρτσκα ακούμε ότι επιθυμούν ε, να επιτύχουν μια, ένα βελούδινο διαζύγιο αυτό όμως δεν προβλέπεται στον Dayton. Κατά τα άλλα, ο πρωθυπουργό της Ρεπούμπλικας Σπέρσκα επιθυμεί ε, να έχει ε, συνεχώς την αυστηρή εφαρμογή της συμφωνίας του Dayton. Στον Dayton όμως δεν αναφέρεται το βελούδινο διαζύγιο. Και εμείς ε, τότε στηρίξαμε τη Συμφωνία Ντέιτον γιατί ήταν η μόνη δυνατότητα να υπάρχει κράτος Βοσνίας-Ερσεγοβίνης. Δυστυχώς όμως η κατάσταση είναι πλέον πολύ δύσκολη και οι πολιτικοί επιτόπου πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν δύο οντότητες, εκ των οποίων η μία θεωρεί ότι είναι κράτος εν κράτη. Όμως ε, Μόνο εφόσον υπάρχει κράτος Βοσνίας-Ερζεγοβίνης μπορούν αυτοί να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βοσνιοκροατική Ομοσπονδία και η Ρεπούμπλικα Σμπέρσκα είναι κομμάτι ενός συνόλου και λειτουργούν μόνο ως σύνολο. Ως εκ τούτου θα πρέπει ε, να χωρηθεί η εξουσία στο κράτος, γιατί αλλιώ το κράτος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό ισχύει σε όλα τα κράτη και όχι μόνο στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση η οποία όπως σας είπα δεν βελτιώθηκε. Το κράτος ε, ακόμα ε, είναι αποδυναμμένο ακριβώς λόγω αυτών των εθνικιστικών κορονών που σας προανέφερα και λόγω του ότι μερικοί δεν επιθυμούν να υποταχθούν σε αυτό το κράτος. Στη Βοστία Σεχοβίνη ακόμα δεν έχουμε ανώτατο δικαστήριο το οποίο να μεριμνήσει για την κατανομή των εξουσιών. Επίσης ε, υπάρχουν συνεχώς επιθέσεις από τη Ρεπούμπλικα Σβέρσκα ε, προς την δικαστική εξουσία. Και όλα αυτά δεν ε, προάγουν την ενότητα. Υπάρχει επίσης μια κατάσταση που γνωρίζουμε όλοι μας. Έχουμε τον ύπατο εκπρόσωπο, τον ανώτατο ύπατο εκπρόσωπο που έχει και μια άλλη ιδιότητα που είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια στιγμή όμως ε, θα μπορούσε να σταματήσει η αρμοδιότητά της, της της εκπροσώπου, γιατί εμείς ελπίζουμε ότι η χώρα θα μπορούσε να δοθεί στα χέρια των υπευθύνων. Τελικά όμως υπάρχει η υπευθυνότητα, μερικοί πολιτικοί δεν αναλαμβάνουν τις ε, ευθύνες τους και μερικοί συμπεριφέρονται ε, σαν ε, η χώρα να θέλει να οδηγηθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως σαν οι πολίτες να έχουν το δικαίωμα να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε ε, ελεύθερο τον δρόμο στην ύπατη εκπρόσωπο. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Την τελευταία φορά όταν ήμασταν στη Βοσνία Σεχοβίνη, αυτό ήταν την άνοιξη αυτού του έτους, διαπιστώσαμε ότι οι πολιτικοί είχαν την θέληση να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις για την ελευθέρωση των ε, θεωρήσεων διαβατηρίων. Και το έκαναν αυτό και πρέπει να τους επενέσουμε, γιατί πράγματι έκαναν ε, κάτι το οποίο το περίμενε οι πολίτες εδώ και πολύ καιρό. Ε, ολοκλήρωσαν και εκπλήρωσαν μάλλον τις προϋποθέσεις του χάρτη πορείας. Θυμάμαι λοιπόν ότι τότε που συζητήσαμε με τους πολιτικούς, μου είπαν οι πολιτικοί, δώστε μας όμω ένα χάρτη πορεία και για άλλα πράγματα. Δεν έχουν καταλάβει ότι Υπάρχει χάρτης πορείας, υπάρχει συμφωνία σύνδεσης, υπάρχουν όλα αυτά που πρέπει να εφαρμοστούν και υπάρχει και ο χάρτης πορείας που έχει σχέση με την ύπατη εκπρόσωπο. Πρόκειται λοιπόν για την ε, ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων. Σε αυτήν εδώ την έκθεση ε, βλέπω κάτι το οποίο πέρυσι με λύπησε, παραδείγματος χάνει το γεγονός ότι στη Βοσνία Ερσεγοβίνη γίνεται λόγος για τις χιλιάδες γυναίκες ε, και τα κορίτσια τα οποία από το 92 μέχρι το 95 βιάστηκαν και κανείς δεν ασχολείται με αυτές. Κανείς δεν τους απέδωσε δικαιοσύνη, ούτε αποζημίωση. Αυτά λοιπόν τα θύματα αντιμετωπίζονται μάλιστα και με έλλειψη σεβασμού και εν μέρη αντιμετωπίζονται και αναξιοπρεπώς. Ούτε προστατεύονται, ούτε στηρίζονται για να φτιάξουν μια καινούργια ζωή. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει ε, να στρέψει την προσοχή της ακριβώς σε αυτό το ένα έστω θέμα και πρέπει τις αρχές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να τις καλέσει και σε σύνολο και μεμονωμένα να αποδώσουν δικαιοσύνη σε αυτές τις γυναίκες. Κατόπιν έχουμε μια κατάσταση στη Βοσνία Ζεγοβίνη που αφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν νομίζω ότι το σύστημα είναι σύγχρονο, δεν ξεπερνάει τις ε, εθνοτικές διαχωριστικές γραμμές και σε πολλές ε, περιπτώσεις δεν ε, είναι στο ύψος ε, των ε, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ένα πρόγραμμα, τη διαβίου μάθηση. Αυτό το πρόγραμμα το ανοίξαμε σε αυτές τις χώρες. Εμείς πιέσαμε την Κομισιόν να ανοίξει αυτό το πρόγραμμα. Από το 2007 υπάρχει αυτό το πρόγραμμα διαβίου μάθησης, ε, ε, έρασμος, κομμένιους, όμως οι χώρες αυτές ε, δεν κάνουν χρήση του προγράμματος και δεν μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος αυτού γιατί υπάρχουν περίπου 13 Υπουργοί Παιδείας. Δεν υπάρχει ένα Εθνικό Υπουργείο Παιδείας που να είναι συνομιλητής της Κομισιόν. Και τα χρήματα τα οποία δίδονται για να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι στο πρόγραμμα αυτό, ε, τα χρήματα αυτά ε, μπορούν να διατεθούν, αλλά όπως σας είπα δεν απορροφώνται. Και αυτό οφείλεται στο ότι η συμφωνία Dayton ε, δεν άλλαξε την κατάσταση που είχε δημορφωθεί από την Ουάσιγκτον δέκα καντόνια με δέκα κυβερνήσεις. Μετά υπάρχει μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση και πάνω από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπάρχει το κράτος. Ε, πώς να λειτουργήσει όλο αυτό. Αυτή λοιπόν την κατάσταση βρήκαμε και στην ε, έκθεσή μας ε, προσπαθούμε να εκφράσουμε τα αιτήματά μας, το τι κατά την άποψή μας πρέπει να γίνει. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι και το Συμβούλιο και η Επιτροπή, κατά την άποψή μου, ε, πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη εξουσία και διπλωματικές ικανότητες. Ο κύριος Μαρτίνος, ο Ισπανός Προεδρεύων και ο κύριος Στάινμπεκ εκ μέρους των Αμερικανών ε, προσπαθούν να έρθουν σε επαφή πέντε μήνες πριν από τις εκλογές, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει σημαντική αλλαγή στο Σύνταγμα. Και το Σύνταγμα πρέπει να αλλάξει αν θέλουμε να λειτουργήσει το κράτος. Ακούμε από την άλλη ότι αυτό κανείς δεν το θέλει, διότι τον προηγούμενο φθινόπερο, όταν προσπάθησαν οι Σουδοί στην Πότμια να επιτύχουν μια συνταγματική αλλαγή, ούτε και αυτοί το κατάφεραν. Και τώρα λένε δεν θέλουμε τίποτα. Εντάξει, δεν ισχύει αυτό για όλους, αλλά ισχύει κυρίως για τον Πρωθυπουργό της Ρεπούμπλικας Μπέρτσκα, που λέει ότι δεν θέλει καμία συνταγματική αλλαγή. Τελεία. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε σε μια κατάσταση η οποία ε, θα επιφέρει στη χώρα δυσάρεστο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς πρέπει να επιδείξουμε μεγαλύτερη σκληρότητα και αυστηρότητα. Σήμερα, διαβάζοντας ότι οι προσπάθειε του κυρίου Μαρτίνο ε, και του κυρίου Στάνμπεκ κατά πάσα πιθανότητα δεν θα οδηγήσουν πουθενά γιατί προετοίμασαν μια δήλωση που κανεί δεν τη δέχεται. Ακούμε ότι ήδη τώρα οι Αμερικανοί λένε μετά τι εκλογέ, εμεί, οι Αμερικανοί θα ε, προωθήσουμε την συνταγματική αλλαγή. Μα πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την τελευταία φορά το 2006 το ίδιο πάλι έγινε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμπεριλήφθηκε καν σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε λοιπόν την ίδια κατάσταση που είχαμε και τότε και νομίζω κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβεί. Κατόπιν υπάρχει το εξή ε, γεγονό. Ε, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο διαπίστωσε, το γνωρίζαμε όλοι, ότι η συμφωνία του Ντέιτον είναι άδικη στο σημείο όπου αναφέρεται ότι ε, στα διάφορα αξιώματα θα πρέπει να εκλέγονται οι πολίτες που προέρχονται από τις τρεις εθνότητες, Βόσνιους, Κροάτες και Σέρβους και οι άλλοι, the others, ε, δεν έχουν ε, καμία ευκαιρία να εκλεγούν. Ποιοι είναι οι άλλοι. Οι άλλοι είναι εκείνοι που δεν μπορούν να πούνε ότι είναι Κροάτες, Σέρβοι ή Μουσουλμάνοι. Όλοι εκείνοι λοιπόν που προέρχονται από ε, μικτούς γάμους, κάποιος ας πούμε που έχει πατέρα Κροάτη και μητέρα από τη Σερβία, τι είναι αυτός τώρα. Αυτός τώρα τι είναι, Σέρβος, είναι Κροάτης αυτός είναι στους others, the others, από αυτούς που δεν μπορούν να εκλεγούν. Αυτό είναι τόσο μειωτικό το να μην ανήκει κανείς στο λαό και να μην έχει εθνότητα να το λένε the others. Και αυτοί οι the others ούτε καν ε, να εκλεγούν δεν μπορούν. Αυτό λοιπόν το ε, διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά την ε, υπόθεση που κινητοποιήθηκε από τον Εβραίο κύριο Σίνσκι. Περιμένουμε λοιπόν μετά τον Οκτώβρη να αλλάξει το στέγμα έτσι ώστε να μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και οι άλλοι, the others. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, πολλές ε, δυσκολίες για να τροποποιηθεί το στέγμα πριν από την εκλογή, από τις εκλογές. Ο κύριος Ντόντιτς προσπαθεί να επιτύχει μία μικρή αλλαγή όπου ε, για το ε, αξίωμα του Προέδρου να μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα ένας από την Ρεπούμπλικα Σφέρτσκα και δύο από την Κροατο-Μουσουλμανική Ομοσπονδία, χωρίς να λέω ότι θα πρέπει να είναι Κροάτης, ε, Σέρβος ή Μουσουλμάνος. Αυτό όμως είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι. Και αν τελικά αυτός είναι ο ελάχιστος κοινό παρονόμαστής, δεν ξέρω κατά πόσον ε, πραγματικά ε, σεβόμαστε, οι πολιτικοί επιτόπου σέβονται την απόφαση του δικαστηρίου. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι επιτέλους πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο δικαστήριο στην Βοσνία Ερσεγοβίνη. Στην γερμανική μετάφραση του κειμένου υπάρχουν ε, γλωσσικά λάθη που δεν θα τα πω εδώ, ε, θα καταθέσω τροπολογίες για να είναι η γερμανική μετάφραση αντίστοιχη της αγγλικής. Επίσης το θέμα της αντιμετώπισης ε, των εγκλημάτων πολέμου, του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, αυτά πρέπει να ληφθούν περισσότερο υπόψη. Επίσης επιθυμούμε ε, στον ποινικό κώδικα να συμπεριληφθεί και η σεξουαλική βία, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να καταβάλλεται αποζημίωση ε, στις γυναίκες και στα κορίτσια που σας ανέφερα προηγουμένως. Γιατί εντωμεταξύ τι γίνεται, ο βιασμός έχει ή αν αναγνωριστεί και έχει αναγνωριστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ε, τότε θα πρέπει να είναι δυνατόν ο βιασμός ε, στη Βοσνία Ερσεγοβίνη να αναγνωρίζεται επίσης και τα κορίτσια, οι γυναίκες ε, που ανέφερα να λάβουν αποζημίωση. Λέμε ότι η επιστροφή ε, των προσφύγων και των εκδιοχθέντων ακόμα δεν μπορεί να είναι ασφαλής, δεν υπάρχουν σχετικές εγγύησεις. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί και το θέμα των καταβλισμών. Θεωρούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν παλαιότερα στη Ρεπούμπλικα Σβέρσκα και οι οποίοι εκδιώχθηκαν στις γειτονικέ περιοχές, γιατί η Ποσαβίνα κοντά στην Πανιαλούκα εξακολουθεί να έχει την ίδια εικόνα όπως ε, και λίγο μετά τον πόλεμο. Και αυτό είναι κρίμα για μια θαυμάσια περιοχή που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Η διαφθορά είναι ένα τεράστιο θέμα και στην κυβέρνηση κατά την ανάθεση ε, δημοσίων έργων, κατά την ε, εκχώρηση των επαγγελματικών αδειών, στην ενέργεια, στις μεταφορές, η διαφθορά. Είναι ένα καθοριστικό θέμα. Και μάλιστα όχι μόνο σε ένα κομμάτι, οριζόντια, σε ολόκληρη την Ομοσπονδία. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτά τα θέματα που αναφέρουμε, κατ' ουσίαν ε, δεν επιθυμούμε να αποδώσουμε ευθύνε μόνο σε μία μεμονωμένη πλευρά, αλλά θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά του και να καταδείξουμε που ε, υπολείπονται πολλά ακόμα. Είπα, το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να προσαρμοστεί σε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα ήθελα να παρακαλέσω να ε, υιοθετήσετε μια δική μου τροπολογία που θα καταθέσω σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση. Γιατί νομίζω ε, παραδείγματο χάρη, ε, στο θέμα των μεών στα νοσοκομεία. Η εκπαίδευση των μεών είναι ανεπαρκής. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε με κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχουμε την αναδιάρθρωση σε αυτόν τον τομέα. Ε, θίγει το θέμα των θεωρήσεων διαβατηρίων. Είδαμε ότι οι πολιτικοί σε αυτόν τον τομέα δούλεψαν καλά και ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, μέσα στην Βοσνία και η ε, μετακίνηση των ατόμων αντιμετωπίζει προβλήματα. Γιατί όσον αφορά τα κοινωνικά συστήματα ε, και τα εργασιακά υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Ε, το να μεταβεί κανείς από το ένα τομέα στον άλλο πρέπει να αντιμετωπίσει ολόκληρους τείχους. Άρα δηλαδή θα πρέπει να μπορεί κανείς να εργάζεται και στη μία και στην άλλη πλευρά. Απαιτούμε επίσης να υπάρξει νομοθεσία σχετικά με την απογραφή του 2011. Βεβαίως εδώ υπάρχουν πρόβλημα γιατί δεν επιθυμούν πολύ να αναφέρεται αυτό που αναφερόταν παλαιότερα ότι δηλαδή θα πρέπει να είναι γνωστό ποιος ανήκει σε ποια εθνότητα. Ο νόμος αυτός ακόμα δεν ε, προετοιμάζεται. Υπάρχει άλλο ένα θέμα, ε, το θέμα της ε, κρατικής ιδιοκτήτησης ιδιοκτησία ε, κράτος είναι η Βοσνία Ερσεγοβίνη. Αλλά η κατανομή της ε, κρατικής περιουσίας είναι ένα σημαντικό κριτήριο και ως εκ τούτου πρέπει να ε, πείσουμε τους πολιτικούς με τον κύριο Σκόντεν, τον, κύριο, τον είπα το εκπρόσωπο, να συνεργαστούν για την κατανομή της ιδιοκτησίας του κράτους. Χαίρομαι που εντωμεταξύ η Ομοσπονδία κατόρθωσε να αποκτήσει κονδύλια γιατί με τον τρόπο αυτό κατόρθωσε και να καταρτήσει νόμους και να πάρει χρήματα από το Διεθνές Νομιωτικό Ταμείο. Είναι καλή και σημαντική και η περιφερειακή συνεργασία. Ε, νομίζω ότι είπα τα περισσότερα, ίσως να και πολλά κενά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την κατανόησή σας. Είμαι πεπισμένος ότι το κάνατε. Έχουμε 11 ομιλητές ε, στο κατάλογο. Το ένα πλεονέκτημα είναι ότι καλύψατε πλήρως την κατάσταση. Οπότε υποθέτω ότι οι ομιλητές θα συντομεύσουν τις παρεμβάσεις τους. Θα δώσω το λόγο πρώτον, πρώτα απ' όλα μάλλον στους σκιώδεις συζητητές και θα ακολουθήσουν οι άλλοι. Εγώ είμαι επικεφαλής αντιπροσωπείας, δεν είμαι σκιώδης. Α, ε, μάλλον σας άλλαξα εγώ θέση, λέει ο πρόεδρος, ε, και σας έκανα σκιώδη ηγητή. Είστε όντως επικεφαλής αντιπροσωπείας. Καταρχάς, ε, να συγχαρώ την επιφανή συνάδελφο, κυρία Πάκ, για μια εξαιρετική έκθεση. Ε, συμπεριέλαβε σχεδόν όλα τα ε, ε, σημαντικά ζητήματα ως προς την κατάσταση που επικρατεί στη Βοσνία. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάποια ζητήματα που πρέπει να τονίσουμε στα πλαίσια αυτού του ψηφίσματος κατά τη γνώμη μου. Αναφέρατε τις εκλογές που θα γίνουν φέτος Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη λένε πολιτικοί παράγοντες ότι δεν είναι σωστός ο χρόνος, τίποτα δεν θα επιτευχθεί, ε, ότι πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια διαφορετική θεώρηση. Το αντίθετο θα πρέπει να θεωρήσουμε την προεκλογική περίοδο ως ε, μοχλό για να ασκήσουμε πίεση στον πολιτικό κόσμο της Βοσνίας ε, για να προβεί σε απαιτούμενες οικονομικές και άλλες μεταρρυθμίσεις. Ε, ίσως να πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν διαφορετική προσέγγιση ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι είναι ουραγός η Βοσνία σε σχέση με γειτονικές χώρες στην οδό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το, αυτό τονίζεται στην έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και από την ε, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη που καλεί επανειλημμένα τους πολιτικούς παράγοντες να κάνουν τα απαιτούμενα βήματα ώστε να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες ε, μεταρρυθμίσεις. Ε, περιορισμένη πρόοδος λοιπόν ως προς τις μεταρρυθμίσεις ε, για εξαιρετικά εκτεταμένη χρονική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί κάποιος να πει ότι η πρόοδος προς την εκπλήρωση των υποσχέσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης ε, σημειώνει εξίσου μεγάλη καθυστέρηση. Πρέπει οπωσδήποτε η χώρα να προχωρήσει με τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στην εγκαθίδρυση ενός πιο συνεκτικού ε, συστήματος ε, και πλέον λειτουργικών ε, δημοσίων υπηρεσιών. Χρειάζονται οικονομικές μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικού κυρίως χαρακτήρα, κατάργηση, σταδιακή κατάργηση όλων των φραγμών για να δημιουργηθεί ένας ενιαίος οικονομικός χώρος και να, αναζωογονηθεί η διαδικασία ιδιωτικοποίηση με τη βοήθεια του ε, προενταξιακού χρηματοδοτικού μέσου ε, ευελπιστούμε ότι θα περατωθούν αυτέ οι οικονομικέ μεταρρυθμίσει. Ε, βέβαια αυξάνεται η ανεργία και πρέπει να το αναφέρουμε γιατί έχει φτάσει στο 40%. Άλλε δύο παρατηρήσεις, Πρόεδρε, θα κάνω. Νομίζω ότι η αναξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ πρέπει, είναι ένα θέμα που πρέπει να αναφερθεί μέσα στο ψήφισμα πρέπει να εξετάσουμε το δεχόμενο συμπερίληψη αυτού του ζητήματος, ε, διότι ε, τα κρατικά ΜΜΕ πρέπει να αναφερθούν διότι συνιστούν σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της ε, μυσαλλοδοξίας για εθνοτικούς λόγους ή άλλους να υπομισθούν τις ευθύνες τους, να ε, λειτουργήσουν προευρωπαϊκά. Τέλος πάντων ίσως είναι ε, ουτοπικό αυτό, αλλά να το αναφέρουμε προτείνω. Κάτι τελευταίο, θέλω να προσθέσω αυτά που πει ε, να εκτιμήσουμε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος για τις θεωρήσεις διαβατηρίων ε, αναμένεται νομοθετικό πακέτο για αυτό το ζήτημα και αναμένεται θετική αξιολόγηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο σύντομα θα επιληθεί του ζητήματο. Ευχαριστούμε ο κύριο Βιγγένιν τώρα που εκπροσωπεί ε, την κυρία Μποσκούτ που είναι σκιώδη εισηγήτρια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Πάκα. Εξ ονόματος ε, της κυρίας Μποσκούτ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε. Ε, ε, έκανε μια εισβάθος ανάλυση η κυρία Πακ και είναι μια έκθεση που έχει ισχυρό έρισμα και δεν χρειάζεται να προσθέσω πολλά πράγματα. Ε, νομίζω θα περάσουν τα σωστά μηνύματα προς τη Βοσνία Ζεγοβίνη αν εγκριθεί το ψήφισμα. Εξ ονόμως της κυρίας Μποσκούτ θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το θέμα των εγκλημάτων πολέμου και των ε, όσων ε, επιβίωσαν ε, γιατί δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής αυτό το ζήτημα μέχρι στιγμής. Για την ομάδα μου, τους σοσιαλιστές, είναι σημαντικό να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για το εξή ζήτημα. Η προοπτική της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας παράγοντας που ενώνει τους ανθρώπους είναι ένα κίνητρο ε, για να γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες λοιπόν. Στις 15 Ιουλίου θα είναι η επέτειος ε, των 15 ετών από την πτώση της Ρεμπέντσα και θα υποβάλουμε και άλλη μια τροπολογία για αυτό το ζήτημα. Κάποια άλλα ζήτημα που ε, θα πρέπει να αναφερθούν τουλάχιστον γιατί είναι σημαντικά η κατάσταση των γυναικών και των μειονοτήτων Εβραίων, ε, Ρώμ, ε, ανθρώπων που έχουν αλλάξει φύλλο. Η Βοσνία Ζεγοβίνη αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα διότι είναι κράτος διέλευσης στην εμπορία ανθρώπων. Κάποιος αναφέρθηκε και στους μετανάστες και σε όσους εσωτερικά έχουν εκτοπιστεί και αυτό πρέπει να αναφερθεί. Επίσης δεν έχει ανοικοδομηθεί και η χώρα από το τέλος του πολέμου. Υπάρχει μεγάλη ενέργεια κυρίως για τους νέους. Πάνω από 40% εμείς ακούσαμε ε, ότι είναι η ανεργία. Ε, ε, αναρωτιέμαι πώς επιβιώνουν οι άνθρωποι εκεί. Κάποια παραοικονομία θα υπάρχει. Είναι νομίζω ένα ζήτημα που πρέπει να αναφέρουμε οπωσδήποτε. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Μέσα από αυτό το ψήφισμα και από την παρουσίαση κυρία ΠΑΚ ε, διαπιστώνουμε την απογοήτευσή σας ε, λόγω της έλλειψης προόδου στη χώρα αυτή. Και θα έπρεπε να αναλύσουμε ίσως, αν, ε, όχι σε αυτό το ψήφισμα, να αναλύσουμε λοιπόν για ποιο λόγο καθυστερεί η πρόοδος, για ποιο λόγο είναι η πρόοδος και όχι ότι εμείς ε, θα επιβάλλουμε τη βούλησή μας, αλλά να βρούμε έναν τρόπο να ε, κάνουμε αυτή τη χώρα να κινηθεί ταχύτερα προς την ε, κατεύθυνση που ξέρει ότι πρέπει να ακολουθήσει για να παραμείνουμε έκπληκτοι που το γνωρίζουν και δεν κάνουν αυτά που πρέπει. Στο Σαράγεβο την περασμένη εβδομάδα οι σοσιαλιστές διοργάνωσαν μια μεγάλη διάσκεψη και ε, αποκομίσαμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια κακοθυμία, ε, δυστημία μάλλον στην περιοχή σχετικά με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εν γέννη στην ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη βλέπουμε τα δέντρα και ξεχνάμε το δάσος, τη συνολική εικόνα δηλαδή. Αυτή είναι πάγια θέση του, της πολιτικής μας ομάδας και ελπίζουμε να μας υποστηρίξει το Κοινοβούλιο ότι δηλαδή η προσχώρηση μέχρι το 2014 ξέρουμε ότι δεν γίνεται μια διεύρυνση στην περιοχή μέχρι τότε αλλά τουλάχιστον να, να φυσίσουμε νέο πνεύμα στη διαδικασία διεύρυνσης και χώρες όπως η Βοσνία Ζεγοβίνη έτσι μπορεί να καταβάλουν νέε προσπάθειε ε, γιατί θα διαπιστώσουν ότι θέλουμε, είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε σκληρά για να ε, προάγουμε την ε, διαδικασία διεύρυνση όχι μόνο για τη Βοσνία αλλά και για άλλε χώρε. Δείτε το νοδικό χάρτη για τις θεωρήσεις, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν σαφείς αιτήσει, ε, στόχοι μετρήσιμοι, ε, μπορούμε να αξιολογήσουμε ε, αμφότερη την διαδικασία. Ελπίζουμε ότι φέτος η Βοσνία θα μπορέσει να τύχει να προσχωρήσει το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης αλλά και η Βοσνία πρέπει να δείξει την αντίστοιχη βούληση και ξαναλέω ίσως ε, αυτό δεν είναι μόνο θέμα αυτού του ψηφίσματος, ως κοινοβουλίο θα πρέπει να κινηθούμε. Ε, Um, and, uh, I... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες που είπαν ότι είναι εξαίρετη η έκθεση της κυρίας Πακ. Πράγματι. Και η παρουσίασή της ήταν πλήρης. Λίγα πράγματα έχω να πω. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που έχει συμπεριλάβει τη μνήα της διαφοράς, το ότι χρειάζεται ανώτατο δικαστήριο, νομική εναρμόνιση, να τονιστούν περισσότερο. Κάποια πράγματα τώρα που θα μπορούσαμε να τονίσουμε περισσότερο και να υπογραμμίσουμε το επίγον πρώτα απ' όλα είναι οι διακρίσεις που γίνονται στα σχολεία. Κάτω από μία σκεπή, μέσα σε ένα σχολείο υπάρχει διάκριση. Είναι απαράδεκτο αυτό μετά το Dayton που ήταν ε, ένα μέτρο προσωρινό. Αλλά κρατάει ακόμα, δυστυχώς. Χαίρομαι που αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη για τα θύματα επίσης και σεξουαλικής βίας, η κυρία Πακ. Ίσως αν τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε δώσει μεγαλύτερη σημασία σε αυτό, ίσως να μην βλέπαμε τους βιασμούς να αποτελούν ε, ένα εργαλείο πολέμου, όπως το βλέπουμε σήμερα στο Κονγκό. Θα έπρεπε αυτό να το είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα. Επίσης θα ήθελα να τονιστεί περισσότερο η ανάγκη μεταρρύθμισης του εκλογικού νόμου. Όπως είπε και η κυρία Πακ το θέμα της διάκρισης που καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Στρασβούργου. Πρέπει να σταματήσει. Έρχομαι τώρα στην ευρύτερη συνταγματική μεταρρύθμιση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν. Ακόμα και αν δεν είναι τόσο ρεαλιστικό ή τόσο επιθυμητό να υπάρξει προθεσμία. Η ημερομηνία δηλαδή καταληκτική. Εγώ μόνο το ανακοινωθέν τύπου της προηγούμενης εβδομάδας διάβασα και φαίνεται ότι η Προεδρία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ε, σχέδιο δήλωσης όπου οι διάφορες πλευρές μετά τις γενικές εκλογές να δεσμεύονται υπέρ της δαγματικής μεταρρύθμισης. Ποια είναι η γνώμη της. Πάντω όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη που υπάρχει για συνταγματική μεταρρύθμιση, προκειμένου να έχουμε ένα κράτος που λειτουργεί, κάτι που είναι προϋπόθεση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, οικονομικές και κοινωνικές ε, πρόοδοι. Μα δεν υπάρχει συμφωνία και υπάρχει ακριβώς αυτή η σύνδεση ανάμεσα στη συνταγματική μεταρρύθμιση και την οικονομική ανάπτυξη γιατί πρέπει να υποφεληθούν από τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζει ότι υπάρχει κάποια πρόοδος όσον αφορά την ελευθέρωση του συστήματος θεωρήσεων εισόδου. Οι αρχές πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, γιατί κάθε φορά που έχουν μπορούν να κάνουν κάτι. τώρα το ψηφίσουμε αυτή την έκθεση, ίσως καλό θα ήταν και να πούμε αν υπάρχει μια θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Πάντως μπορούμε να συγχαρούμε την Φωσνία που έγινε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως ε, χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου. Και καλό θα ήταν να μιλήσουμε και για το ψήφισμα για την ε, Σερβενίτσα από πλευράς της Σερβίας. Ακόμα και αν έχει αποφύγει τον όρο γενοκτονία. Καλό είναι που αν μη τι άλλο αναγνωρίζεται και η, εκαιρότητα, η και να ενθαρρύνουμε τον, ε, το Βοσνιακό Κοινοβούλιο να εγκρίνει επίσης ένα ψήφισμα από τη δικιά τους πλευρά. Τέλος, Υπάρχει ένα σχέδιο για περιφερειακή διάσκεψη στο Σαράγεβο 1η Ιουνίου όσον αφορά την πρόοδο για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ήμουν το Μάρτιο στην περιοχή, δεν πήγαν ηγέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή εκπροσωπιόταν το Κοσυφοπέδιο. Ελπίζω να μην έχει προηγηθεί κάποια συμφωνία με τη Σερβία, που δεν θα ήταν αποδεκτό. 1η Ιουνίου ελπίζω να υπάρξει, ό,τι και να κάνει η Σερβία, να υπάρξει εκπροσώπηση πλήρης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι θλιβερό να ακούμε ότι μια χώρα η οποία τελικά που θέλει να έχει καλές σχέσεις με τους γειτονές της, ότι η ίδια απομονώνεται κατά κάποιο τρόπο και περιορίζεται. Και για να μπορέσουμε αυτό να το ξεπεράσουμε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλουμε σταθερότητα στην περιοχή, καλό θα ήταν να διακανονιστούν τα πράγματα μια για πάντα. Και είναι θλιβερό τα παιδιά που πάνε σχολείο, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, στην πρόσβασή τους ακόμα το μπορεί που πάνε σχολείο, υποφεύγουν από το σχολείο. Συγχαίρω την ε, εισηγήτρια πάντως για την έκθεσή της. Χαίρομαι που αναφέρει την βία σε βάρος των γυναικών, τους βιασμούς και εκτός πολέμου. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτό θέλουμε να αλλάξει. Τώρα η θέση των μειονοτήτων στη Βοσνία. Μιλήσαμε για τα παιδιά που χωρίζονται όταν πηγαίνουν στο σχολείο και το ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι άλλοι οι άλλοι, όπως και οι δημοκράτες και εμείς θέλουμε να μην αναφέρονται οι άλλοι σαν να πρόκειται για μια άλλη εθνότητα ή για μια άλλη θρησκεία, είναι αυτοί που προέρχονται από μικτές οικογένειες. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω την Επιτροπή, γιατί η κυρία Πακ μιλάει θετικά για την ρύθμιση όσον αφορά την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Η προθεσμία όμως, καλοκαίρι του 2010, φτάνει όπου να είναι. Οπότε, τι θα γίνει. Θα γίνει κάτι. Η Βοσνία Αρζεγοβίνη, ακούσαμε πώς έχω προχωρήσει. Η Κομισιόν έχει προχωρήσει αρκετά. Εγώ φοβάμαι πως όχι. Και μια άλλη ερώτηση που πρέπει να θέσουμε στους αυτούς μας είναι η Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλό να συνδυαστεί με τον υπατό εκπρόσωπο. Είναι καλή ιδέα κάτι τέτοιο. Να συνδυαστεί δηλαδή η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση της Βοσνίας Ερσεγοβίνης με μια άλλη πλευρά. Τι μπορούμε να κάνουμε. Τέλος, οι πράσινοι θέλουν να τονίσουν και το θέμα της αηφόρου ενέργειας. Η Βοσνία χρειάζεται βοήθεια. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη, για να το πω πιο σωστά, χρειάζεται βοήθεια και μια στρατηγική για το ενεργειακό. Είναι καλό που γίνεται κάτι, που υπάρχουν ε, υδροελεκτρικά εργοστάσια. Είναι καλό. Πρέπει να γίνουν πάντως περισσότερα και να βοηθηθεί περισσότερο η χώρα όσον αφορά το ενεργειακό της ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και η κυρία Κοπά και η κυρία Ιμπρουζίτς μετά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Πακ για την έκθεσή της και να ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση. Παρόλο που οι επισημάνσεις της και η κριτική της είναι σωστές και η απογοήτευσή της είναι απολύτως δικαιολογημένη, διατηρώ σοβαρές αμφιβολίες για αν η υψηλή και καταγγελτική τόνη που υιοθετεί το κείμενο είναι κατάλληλη. Ίσως φανεί υπερβολικό, αλλά ας μου συγχωρεθεί η υπερβολή. Ε, κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφασίσει αν απευθύνεται σε ανεξάρτητο κράτος ή σε προτεκτοράτο. Αν συμφωνούμε ότι η Βοσνία είναι ανεξάρτητο κράτος που έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ύφο της έκθεσης κατά τη γνώμη μου δεν είναι παραγωγικό. Παράλληλα, θα περίμενα και μια νότα αυτοκριτικής από μεριάς της Ένωσης για επιλογές που επέτειναν τα διέξοδα. Φυσικά και πρέπει να προχωρήσει η συνταγματική μεταρρύθμιση. Όλοι γνωρίζουμε, και το ανέφερε η κυρία Πακ, ότι το Dayton ήταν ο ενδεδειγμένος τρόπος για να σταματήσει η αιματοχυσία. Όμως, η δογματική προσήλωση για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτό οδήγησε στην πλήρη εθνικοποίηση όλων των διαφορών στη χώρα. Και είναι γνωστό ότι αν δεν ανήκει σε μια εθνική ομάδα δεν υπάρχει σαν πολίτης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ε, δεν θα μπω σε συγκεκριμένα θέματα, θα σημειώσω μόνο δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα, με τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή έχουμε, είναι κατά τη γνώμη μου μη ρεαλιστική αναφορά στην απελευθέρωση των θεωρήσεων πριν το καλοκαίρι. Μακάρι να μπορούσε να συμβεί, σαν κοινοβούλιο το στηρίξαμε, αλλά δεν έχει νόημα να καλλιεργούμε προσδοκίες οι οποίες δεν φαίνεται να μπορούν να ελοπίθουν. Δεύτερο σημείο, ε, το ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι, ότι χρειάζεται κάποια αναφορά στις εκλογές του Οκτώβρη του 2010. Για τα υπόλοιπα θα κατατεθούν τροπολογίες και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ε, ξέρετε το μειονέκτημα όταν ε, παίρνει κάποιος το λόγο προς το, το τέλος του καταλόγου είναι ότι δεν έχει και πιέζεται πολύ από το χρόνο. Τέλος πάντων, θέλω να συγχαρώ την κυρία Πακ ε, για το σχέδιο του ψηφίσματος που συνέταξε. Υπάρχουν ε, κάποια πραγματάκια που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και να βελτιώσουμε το κείμενο, αλλά εγώ δεν θα μπω στον πειρασμό γιατί ε, καλύπτονται πάρα πολλά ζητήματα. Ε, το θέμα των ανοικίων μεταρρυθμίσεων, τη σχέση της Βοσνίας της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, των ελλείψεων που υπάρχει, υπάρχουν συγγνώμη, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στον τομέα της υγείας. Τέλος πάντων, τα σημαντικότερα ζητήματα καλύπτονται και θα μπορούσα να ακολουθήσω κάποιες ε, προτάσεις ε, συναδέλφων ε, για το θέμα των ΡΟΜ, παραδείγματος χάρη. Θα υποβάλω τροπολογίες, δεν θα το σχολιάζω τώρα. Ήθελα να πω μόνο κάτι. Ακούσαμε επανειλημμένα αναφέρονται δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι η Βοσνία Ριζεγοβίνη είναι μια χώρα που συνιστά χώρα διέλευσης ε, για την εμπορία ανθρώπων. Και δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες ε, και είχα καταλάβει ότι δεν υπάρχει υποστήριξη και γι' αυτό δεν συμπεριλείπει το ζήτημα μέσα στο σχέδιο ψηφίσματος, αλλά το άκουσα από τους συναδέλφους ε, και άρα δεν ισχύει αυτό. Και υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες Και ε, ξέρετε ότι δεν αληθεύουν πάντοτε και ορισμένες ε, χώρες που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί η καταστήση είναι χειρότερη από την Βοσνία Ζεγοβίνη. Δεν είναι τα πράγματα που θέλουμε να τα παρουσιάσουμε. Επίσης ο κύριος Αργεντίνη τι μας είπε. Ε, μας μίλησε για το γραφείο του είπα του εκπροσώπου ότι ταυτίζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται. Εμείς ε, έχουμε κάποιον ε, που έχει... Έχουμε τον ύπατο εκπρόσωπο και τον ειδικό απεσταλμένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ειδικό απεσταλμένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο ύπατο εκπρόσωπο συνδέεται με τη διεθνή κοινότητα. Και αυτή η διάκριση, αυτή η διαφορά οδήγησε στη συζητήση σχετικά με το αν και πότε ε, θα κλείσουμε το γραφείο του υπάτου εκπροσώπου. Και θέλω να υποστηρίξω τη θέση της Ντόρης. Δεν πρέπει πρόωρα να το κλείσουμε το γραφείο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση. Γιατί Μόνο έτσι εκείνοι οι εθνικιστές θα αναγκαστούν να κάτσουν στο τραπέζι και να διαπραγματευτούν. Επίσης, η κυρία Κοπά πολύ σωστά το έθεσε το ζήτημα. Τι μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. είναι αιτιολογημένο να εξηγήσουμε για ποιου λόγου οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση και να δούμε τι γίνεται με αυτή τη διπλή εθνικιστική, ε, με αυτή τη διτή ηθαγένεια. δεν υπήρχε τιμότητα να δράσουμε με πυγμή εξ αρχής. Γι' αυτό οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Εμείς την προκαλέσαμε την κατάσταση στο Dayton, στη συμφωνία Dayton, είχαμε προβλέψει ότι θα στείλαμε κάποιον, αλλά επίσης ε, ε, θέλαμε να επιτύχουμε την εναρμόνιση και θέλαμε να ε, οι συνομιλητές μας ε, να, μπορεί να συμμετάσχει στο διάλογο και να ε, ε, μπορούμε να συνομιλήσουμε και με τις μειονότητες. Και η δημοκρατία της Σερβίας συνέχεια λειτουργούσε ως τροχοπέδι στη διαδικασία και το είδαμε επανειλημμένα και δεν πιστεύω ότι παρά είναι ε, σκληρή η Ντόρις σε αυτά που λέει. Πρώτη φορά λέμε τα, τα πράγματα με το όνομά τους. Πρώτη φορά ε, τοποθετούμαστε και κατακρίνουμε αυτό που έχει συμβεί και αυτό που δεν έπρεπε πριν από 15 χρόνια εμείς να επιτρέψουμε να συμβεί. Τα υποβάλλω σχετικέ ε, τροπολογίε. Ε, θα ζητήσω από του συναδέλφου να υποστηρίξουν το κείμενο ω έχει. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάτσιν, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο, την κυρία Πακ, για το ψήφισμα. Είναι πληρέστατο, ρεαλιστικότερο, ε, ρεαλιστικότατο συγγνώμη, και εξισορροπημένο το ψήφισμα είναι ακριβές και μπορεί να αποτελεί σωστό έρισμα, σωστή βάση για τις μελλοντικές μας εργασίες. Θα υποβάλουμε πάντως κάποιες τροπολογίες για να δείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα μέσα στο ψήφισμα. Ευχαριστούμε την κυρία Πακ που αναφέρθηκε στα θύματα, κυρίως τα, τις γυναίκες θύματα του πολέμου στη Βοσνία. Δίκιο έχει συναδελφός μου. Οφείλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο ζήτημα των γυναικών που ήταν θύματα αλλά μην ξεχνάτε και ότι οι πέτοι για αυτά τα εγκλήματα φεύγουν από τη Βοσνία. Εγώ γνωρίζω μια οικογένεια που έπεσε θύμα βιασμού και τώρα μένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον ίδιο δρόμο με τον αυτούργο που πήρε άσυλο σε αυτή τη χώρα. Ε, καταλαβαίνετε το δράμα αυτής της οικογένειας. Και αυτή η χώρα που χορήγησε το άσυλο ισχυρίστηκε ότι είναι παλιός ο βιασμός ε, και έχει παραγραφεί. Δεν γίνεται δίωξη. Και άρα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρότερα το ζήτημα και να έχει χρυσή ευκαιρία να ε, αναφερθούμε τουλάχιστον στο ζήτημα. Για τη Στρεμπρένιτσα τώρα. Πολλοί στη Βοσνία, ναι, δεν εγκρίνουν το ψήφισμα και είχα και εγώ απευθύνει επικρίσεις για το ψήφισμα αυτό για τη Σερβία, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι καλό γιατί το ζήτημα της Βοσνίας πρέπει να το με σοβαρότητα και το ίδιο και τη Σερβία. Η Βοσνία Ζεγοβίνη μόνη της θα πρέπει να χαράξει το δρόμο της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και όντως πιστεύω ότι δεν έχει σημειωθεί ταχεία πρόοδος. Είναι Παναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια είναι παλιά η ιστορία. Πολλοί πολιτικοί στη Βοσνία ε, κάνουν επιμελείς δηλώσεις. Άλλοι θεωρούν ότι σε αυτό το ε, τελευταίο στάδιο πρέπει να ε, αποσυντεθεί η Βοσνία για να λυθεί το πρόβλημα. Άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να αποσυνδεθεί η Σερβία. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι δεν είναι βιώσιμη αυτή η λύση. Ε, τα θύματα της πολιτικής, ξέρετε ποια θα είναι, η οικονομία. Τι θα γίνει αν οι επενδυτές ε, δεν προτίθενται πλέον να επενδύσουν στη χώρα. Ε, σίγουρα δεν θα είναι επωφελές ένα τέτοιο μέτρο για την οικονομία και άρα ε, πιστεύω ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου και το Κοινοβουλίου, θα έπρεπε να ε, προτείνουν μια διαφορετική προσέγγιση, να ενθαρρύνουμε δηλαδή μια νέα θετική, δεσμευτική, συνενετική προσέγγιση ε, που θα προετοιμάσει τη Βοσνία για το επόμενο βήμα ε, ε, στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ταχεία όμως η πρόοδος, είναι ουραγός, είπαμε, η Βοσνία σε σχέση με άλλες βαλκανικές χώρες, αλλά δεν φταίνε οι πολίτες. Παρ' όλα αυτά, εκείνοι εξέλεξαν την πολιτική ελίτ που σαφώς κατέδειξε στην τωρινή θητεία της ότι δεν ε, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις ε, προκλήσεις ε, που πρέπει να αντιμετωπίσει η Βοσνία για να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιάσκο Φίντσι, αυτή η περίπτωση, τι έγινε. Δεν υπάρχει υπαρκής πολιτική βούληση για να εφαρμοστεί η απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Τι πρέπει να γίνει είναι να ε, διοργανωθούν νέες εκλογές στη Βοσνία, να ε, ανακηρυχθεί ο νέος πρόεδρος, είπαν κάποιοι. Είστε σίγουροι ότι θα υπάρξει, θα οριστεί η ημερομηνία προσχώρησης ε, για τη Βοσνία εάν δεν μπορούν όλοι οι πολίτες ισότιμα να ψηφίσουν ή να, εκλέξουν να εκλεγούν. Είναι ασυγχώρητο από πλευράς μας, πιστεύω εγώ, να υποχωρήσουμε τώρα. Τώρα πρέπει να αγωνιστούμε για να μεταρρυθμιστεί ο εκλογικός νόμος. Μόνο έτσι μπορούμε να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Αλλιώς θα περιμένουμε άλλα τέσσερα χρόνια για να ορίσουμε ημερομηνία προσχώρησης για τη Βοσνία. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να ε, περάσουμε για την Βοσνία. Δεν θα μιλήσω τώρα για τις θεωρίες και την απαλλαγή κτλ. Τα, λοιπά. τα είπαν οι συνάδελφοι. Για τα ε, επόμενα στάδια πάντως μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα και θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες ε, που πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουν το ψήφισμα. Πάντως το, ε, το ψήφισμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μελλοντικές εξελίξεις στη Βοσνία. Uh, έχουμε λοιπόν άλλους τρεις ε, ομιλητές εκτός από τον κύριο Μίλαν που είναι ε, διευθυντής στην ε, μετά η κυρία Πάκ και έχουμε και άλλο θέμα. Και ας μην ξεχνάμε και το ρολόι. Θα ήθελα να ε, δώσω το λόγο στον κύριο Πόσελτ, μετά στον κύριο Σβόμποντα, στον κύριο Πρέντα, Μιρέλ και Πακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι περιμέναμε τόσο καλή δουλειά από την εισηγήτρια, αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα από τη συζήτηση που πρέπει να τα επισημάνω. Εγώ σας ε, προειδοποιώ, δεν θα πρέπει επουδενή να αμφισβητηθούν τα δύο αξιώματα των ύπατων αρμοστών. Η έκθεση ε, πρέπει να δώσει ευκρινές μήνυμα για την ενίσχυση ε, των δύο ύπατων εκπροσώπων. Ε, θα χρειαστεί να παραμείνουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και επίσης και τα άτομα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη υποστήριξη εκ μέρους μας. Έχουμε και ένα θαυμάσιο άνθρωπο και έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος αυτός δεν στηρίζεται επαρκώς από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω στο σχέδιο ένα σημείο που αναφέρει ότι ε, πρέπει να ασκηθεί κριτική και στους δικούς μας τους ε, θεσμούς. Οι θεσμοί αυτοί οφείλουν να επιδείξουν περισσότερες ηγετικές ικανότητες. Νομίζω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό ε, μπορούμε και να άρουμε τις επιφυλάξεις της αδέλφου Κοπά που δεν είναι πια στην αίθουσα. Είναι σημαντικό να τοποθετηθούμε με σαφήνεια στους πολιτικά υπεύθυνους ε, στη χώρα. Αυτό όμως θα το κατορθώσουμε μόνο εφόσον ε, μιλήσουμε ειλικρινά και με τη διεθνή κοινότητα η οποία φέρει ευθύνη για την αθλειότητα. Ε, συνταγματική μεταρρύθμιση. Γιατί δεν προχωράει τίποτα στη Βοσνία τη Γιατί ε, η συμφωνία του Dayton έχει αποτύχει και διότι η χώρα με τις δικές της και μόνο δυνάμεις δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτό το ε, λάθος μόρφωμα. Ε, λέγοντας λοιπόν ότι οι άνθρωποι επιτόπου πρέπει να αλλάξουν την κατάσταση, αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Εμείς οφείλουμε να συμμετάσχουμε ενεργά και όσο σημαντικό και αν είναι ε, να αναζητούμε την κοινωνία των πολιτών. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι αν δεν υπάρχει το εθνοτικό στοιχείο στο Σύνταγμα δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόοδος. Και η Βοσνία Σεγοβίνη θα προοδεύσει μόνο εφόσον βεβαίως και υπάρχει η κοινωνία των πολιτών και ενισχυθεί το κεντρικό κράτος, αφετέρου όμως εάν υπάρχει ένα κράτος τριών μικρότερων ισότιμων κρατών, ε, δηλαδή Βοσνίων, Μουσουλμάνων, Κροάτων και Σέρβων. Και Κροάτες δεν εννοώ μόνο τους Ερζεγοβίνιους, αλλά και τους ε, ε, κεντρικά Βόσνιους που έχουν καταταλαιπωρηθεί, αναφέρθηκε ήδη η Σαβίνα το να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, αυτό θα είναι το μεγάλο καθήκον μας κατά τα επόμενα χρόνια. Και αν δεν το κατορθώσουμε αυτό, τότε θα είμαστε εδώ ακόμα 10-20 χρόνια και θα διαμαρτυρόμαστε και τότε ότι δεν έχουν λάβει χώρα οι μεταρρυθμίσεις. Ο κύριος Σβόμποντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προφανώς η έκθεση της συναδέλφου κυρίας Πάκ είναι μια πολύ καλή έκθεση. Εγώ δεν θέλω να πω μόνο, δεν να πω που συμφωνώ, μόνο τα σημεία εκείνα όπου έχω λιγάκι διαφορετική άποψη. Συμφωνώ και δεν κατανοώ γιατί λίγο πριν από τις εκλογές ε, οι Μορατίνους και οι Στάνμπεκ αρχίζουν να λένε πάλι τα ίδια. Τους έχουμε κάθε επιτυχία. Πρέπει ε, τα πράγματα που μπορούμε να πετύχουμε να τα επιδιώξουμε. Και όσον αφορά ε, το θέμα της ε, εθνότητας. Εγώ άκουσα ότι η Ρεπούμπλικα Σέρψκα είναι πρόθυμη να κάνει περισσότερα για τον πρόεδρο. Αλλά όταν υπάρχει πρόοδος πρέπει και να υλοποιηθεί αυτή. Και πρέπει να πάρει κανείς ε, τα πράγματα όπως τούρχονται. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που βλέπω να υπάρχει. Δεύτερον, είπα τους εκπρόσωπος. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι λιγάκι υπερβολικό. Αυτή η υπερβολική υποστήριξη σήμερα δεν μας επιφέρει τίποτα. Ας είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει αυτός εδώ και χρόνια και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ε, η εξουσία δεν αρκεί αν δεν θέλουν οι άνθρωποι. Εντάξει, πρέπει να το δεχτώ. Αυτό όμως που δεν δέχομαι είναι ότι ο ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναφέρεται καν. Για μένα όμως αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί ο δικός μας ο, ο συνομιλητής είναι ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατανοώ βέβαια το ότι η κυρία Πάκ δεν θέλει να το θίξει το θέμα, αλλά υπάρχει κάτι που είναι πολύ δύσκολο για την κυρία Άστον. Δηλαδή, έχει νόημα τώρα τον ε, ειδικό εκπρόσωπο να τον κάνει επικεφαλής αντιπροσωπείας ή αυτός ε, να παραμείνει με το... Ε, δικό το γραφείο και μετά να γίνει συνένωση των ε, δύο αξιωμάτων, των δύο γραφείων αν θέλετε. Πάντως ε, ο θεσμός ως ε, ειδικό απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όταν μιλάμε για την υπατή εκπρόσωπο, εμείς αυτό πρέπει να το στηρίξουμε. Και για να μην υπάρχει καμία ε, παρεξήγηση, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος ε, Πόσελτ ε, σε αυτό το θέμα, ότι έχουμε έναν πολύ καλό εκπρόσωπο, όχι μόνο γιατί είναι αυστριακός, είναι πολύ καλός, αλλά εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το ότι είναι εκπρόσωπος ειδικό απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πόσελτ, εάν τώρα αρχίσουμε από εδώ να ε, προσπαθούμε να ανατάξουμε την ε, Βοσνία Τσεκοβίνη. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε τις ε, προϋποθέσεις για λύση στην Βοσνία Ερσεγοβίνη. Πρέπει να δουλέψουμε με τις διοντότητες που υπάρχουν και να δούμε και οι Κροάτες να πάρουν τα απαραίτητα δικαιώματα. Τέλος, εγώ δεν συμφωνώ με το 7 και το 6 αλλά κυρίως με το 7. Δεν είναι μόνο η Ρεπούμπλικα Σέρψκα δεν είναι μόνο η Ρεπούμπλικα Σέρψκα, αλλά και άλλοι που έχουν πει πράγματα ε, που δεν είναι ικανοποιητικά. Και όταν λέμε στο 7 ότι καλούμε όλους να δεχθούν τη συμφωνία του Ντέιτον στο σύνολό της ή να την αλλάξουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει ένα λειτουργούν κράτος, ε, ε, με αυτό συμφωνώ. Δεν συμφωνώ όμως ούτε με τον κύριο Ντούντικ, ούτε με τον κύριο που λέει ότι πρέπει να φύγουν οι εθνότητες. Γι' αυτό λοιπόν ε, στην παράγραφο 7 θέλω να δώσω ένα σαφές μήνυμα και στις δύο πλευρές. Ε, δώστε στον Dayton μία ευκαιρία. Αυτή είναι η προϋπόθεση έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να έχουμε πρόοδο. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ την κυρία Πακ. Ε, δύο σύντομες ερωτήσεις θα κάνω. Ε, πρώτα απ' όλα χαίρομαι που είναι σαφέστατο το σημείο 12 του ψηφίσματος για την ε, πραγματικά αναγκαία ε, τροποποίηση του συντάγματος. Επίσης, ε, η τήρηση ε, της ε, σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητη για τις κρατικές δομές. Η κυρία Κοπάνα ρωτήθηκε, είναι κράτος προτεκτοράτο, η Βοσνία τι είναι. Γι' αυτό χρειάζεται αναθεώρηση του συντάγματος ε, για να ε, διευκρινίσουμε την εθνική ταυτότητα και μην ξεχνάτε και την απόφαση του δικαστηρίου στο Στρασβούργο. Ο Πρωθυπουργός ε, της ε, Δημοκρατίας Περσέρφσκα, μίλησε, ε, προώθησε την ε, ιδέα να μποϊκοτάρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι νομίζαμε ότι ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο, αλλά δεν ήταν. Φανταστείτε να βγαίνουν τέτοια λόγια από το στόμα του Πρωθυπουργού πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες και θα υποβάλω σχετική τροπολογία. Πρόεδρος, ε, ε, ο κύριος ο διευθυντής για τις ΔΕΛΤΑ Διεύρυνση, θα πάρει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Πάκη για, την για το εξαιρετικό ψήφισμα που συνέταξε. Συμφωνώ με την κρίση της για την κατάσταση στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Έχει επιδεινωθεί το τελευταίο μήνα η κατάσταση και προχωρούν πολύ αργά οι μεταρρυθμίσεις και η οικονομική κρίση δυσχεραίνει περαιτέρω τα πράγματα. Το 2010 είναι έτος εκλογών και άρα ε, θα επιδεινωθεί περαιτέρω ε, η κατάσταση και εδώ και κάποιες εβδομάδες Έχουμε ακούσει ε, κάποιους ε, ε πύρινους ε, λόγους ε, στη Βοσνία και σίγουρα θα συνεχιστεί αυτό και θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Με ο ύπατος εκπρόσωπος ή ύπατη εκπρόσωπος και ο, ε, Επίτροπος Φιλέ επισκέφθηκαν την Βοσνία για να μιλήσουν για το δημοκρατικό μέλλον της χώρας και για να καλέσουν τους ηγέτες και τις νέες αρχές γιατί μόλις είχε ορκιστεί η νέα κυβέρνηση να μεριμνήσουν ούτως ώστε ε, τα ερχόμενα δύο χρόνια να οδεύσει προς την Ένωση η Βοσνία. Αυτός είναι ο κοινό μας στόχος. Για να υλοποιηθεί ε, πρέπει να καταβάλουν τι απαιτούμενε προσπάθειε ε, οι ηγέτε τη Βοσνία. Προ το παρόν δεν έχουν κάνει πολλά πράγματα. Τι πρέπει να κάνουν. Πρώτα απ' όλα τι συνταγματικέ μεταρρυθμίσει. Έγινε μια σοβαρή απόπειρα πέρσι το φθινόπωρο. Ίσως είναι και το μοναδικό σημείο που δεν συμφωνώ 100% με την κυρία Πακ η Σουηδική Προεδρία μαζί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από κοινού με τη ΣΥΠΑ ε, κατέβαλαν ε, προσπάθεια για να θέσουν επιτάπητο στο ζήτημα των ε, ελαχίστων αλλαγών για το τροποποίησεων μάλλον του συντάγματο. δεν ήταν εξαιρετικά φιλόδοξο, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάπως λειτουργικό. Και δεύτερον, και αυτό είναι σημαντικό, και η κυρία Πάκα και διάφοροι ε, συνάδελφοί της θα το ανέφεραν στη συζήτηση. Πρέπει το Σύνταγμα να ευθυγραμμιστεί με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μετά από την απόφαση και του Δεκεμβρίου. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη ε, βαρύτητα. Ε, αλλά ε, δεν ναι, τελεσφόρησαν οι προσπάθειες. Παρόλα αυτά υπήρξε αυτή η δέσμευση και τώρα υπάρχουν διάφορες εναλλακτικέ λύσεις για τους ηθήνοντες στη Βοσνία για να επομεστούν τις ευθύνες τους και να ευελπιστούμε, τροποποιήσουν το Σύνταγμα πριν τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργό έχει δρομολογήσει και ένα σχέδιο δράση πριν από κάνα δύο εβδομάδε. Ελπίζουμε ότι θα ε, στεφθεί με επιτυχία. Ε, βέβαια, αυτές τις μέρες δεν είμαστε και τόσο αισιόδοξοι, ήδη έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις ε, και ε, δεν υπάρχει πάντοτε η αναγκαία πολιτική ε, βούληση, μόνο σποραδικά. Και ενώ επιθυμεί σφόδρα η χώρα να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διοργανώσει δεύτερη φορά εκλογές και εξακολουθούν κάποιοι πολίτες να μην μπορούν να εκλεγούν ούτε στο Κοινοβούλιο, ούτε να καταλάβουν αξιώματα στην Προεδρία. Άρα, παραβιάζει τη διμερή συμφωνία το άρθρο 2 η χώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα ε, και άρα έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Πακ όταν λέει πως ε, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, γιατί το να προσχωρεί κάποιος στην Ένωση μην ότι και τις αξίες της. Ε, ε, πριν από λίγες μέρες ε, συναντηθήκαμε με βουλευτές ε, στο Σεράγιβο και με ευρωβουλευτές για να εξηγήσουμε και πάλι τι πρέπει να γίνει και να προσαρμοστεί ο νόμος για την απογραφή. Ελπίζουμε να σημειωθεί επιτυχία. Συνεχίζουμε τον τακτικό διάλογο με τις αρχές μετά την ε, υπογραφή της ε, συμφωνίας. Ε, Σε, συνεχίζουμε με τις αρμόδιες υποεπιτροπές. αυτό... Έχει ήδη προσυπογραφεί από 20 χώρες, θα αρχίσει από τον Ιούνιο, πρέπει να θεσπιστεί ε, ε, ο θεσμός της κρατικής επιχορήγησης για την SA, αλλά ε, και ενώ έχει σημειωθεί πρόοδο σε άλλες ε, χώρε, ε, στη Βοσνία υπάρχουν καθυστερήσει. Η μόνη εξαίρεση είναι οι θεωρήσεις. Του τελευταίου μήνε σημειώθηκε πρόοδο. Για ποιο λόγο να ρωτιόμαστε, γιατί οι πολιτικοί ίσω ίσως δεν τολμούν να δώσουν την εντύπωση ότι δεν κάνουν τα πάντα για τους πολίτες τους. Ίσως αυτός είναι ο λόγος, τέλος πάντων θετικό είναι. Ε, και αυτό καταδεικνύει ότι μπορούμε να ε, επιτύχουμε πολιτική συνένεση και τότε θα έχουμε απτά αποτελέσματα. Ε, λάβαμε παρατηρήσεις των αρχών και θα ολοκληρώνουμε τώρα την αξιολόγησή μας και ε, είμαι σίγουρος ότι σύντομα, σύντομα θα υποβάλουμε σχετική πρόταση. Να πω κάτι τελευταίο για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Είναι σημείο κλειδί όντως, όντως. Είναι πολύ σημαντικό, είναι απαραίτητο ε, να απελευθερωθεί το καθεστώς για τις ε, θεωρήσεις για τους πολίτες της Βοσνίας της Ζεγοβίνης. Αλλά είναι σοβαρό το ζήτημα και για τα κράτη-μέλη οι οδικοί χάρτες για την απαλλαγή είναι ε, ίδιοι για όλες τις χώρες. Ακολουθούμε την ίδια μεθοδολογία, την ίδια προσέγγιση για όλους. Και θα ήθελα να πω ε, ανοιχτά ότι δεν μπορεί κανείς να το καταλογεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, να καταλογεί δηλαδή στην Επιτροπή αυτό που το Συμβούλιο δεν μπορούσε να καταφέρει πέρσι όταν οι άλλες τρει χώρες που τελικά ε, εισήλθαν στο καθεστώς απαλλαγή, ε, δεν τα κατάφερναν. Δηλαδή η Βοσνία σήμερα θα μπορούσε να έχει απαλλαγή από τις θεωρήσεις αν είχαν εργαστεί καλά οι αρχές της Βοσνίας όταν γινόταν οι διαπραγματεύσεις. Δεν μπορείτε να μας το καταλαγίζετε και ε, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια που χρειάζεται για να ε, επέλθει απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, αλλά έχουμε καθυστερήσει. Όπως και η κυρία Πακ, ε, ε, λυπούμεθα και εμείς, διότι έχουν διωχθεί ε, ολιγάριθμα εγκλήματα πολέμου, κυρίως όταν μιλάμε για σεξουαλική κακοποίηση. Και η διεθνή στρατηγική για τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να ενισχυθεί, τουλάχιστον. Έχει, έχουν έχει εγκριθεί σχέδιο δράσης, αλλά δεν έχουν εγκριθεί ακόμη οι νόμοι και οι νομίσκοι που χρειάζονται για να εφαρμοστεί η συμφωνία. Ε, και ε, η αρχική ημερομηνία ήταν το 2010. Εμείς τώρα έχουμε ζητήσει αξιολόγηση της μεταρρύθμισης, αξιολόγηση πριν να λάβουμε δέσμευση το 2011, τόσο ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων για μια μεταρρύθμιση, για την οποία όμως δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μας πραγματική ουσιαστική πολιτική βούληση από πλευρά των αρχών της Βοσνίας Εζεγοβίνης να πάρουν σωστέ αποφάσεις. Επίσης θα συμφωνήσω ότι είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με την κοινωνία των πολιτών η UHR στην, ε, με την βοήθειά μας ε, έχει ένα εκτενές ε, πρόγραμμα όπου γίνονται συναντήσεις με βουλευτές και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό και επίσης υπάρχει άμεση συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Υπάρχουν πολλά υποσχόμενες νέες μη κυβερνητικές οργανώσεις στη Σερβία και στην Κροατία υπάρχει και η πρωτοβουλία για την αλήθεια και για την ε, συμφιλίωση για να αντιμετωπίσουμε το πρόσφατο παρελθόν ε, και ε, πραγματικά είναι σημαντική με τέτοια πρωτοβουλία. Θα συμβούσα και με τον κύριο Κούκαν για την ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αυτό πρέπει να αναφερθεί στο ψήφισμα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που ήγηραν οι ομιλητές ε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, τέλος πάντων για την πλειοψηφία τους θα συμφωνήσουμε. Τέλος, ε, θα ήθελα να συμφωνήσω και πάλι με την κυρία Πακ ε, για το σύστημα των δύο σχολείων υπό την ίδια στέγη. Είναι απαράδεκτο προετοιμάζει γενναίες που στην καλύτερη περίπτωση θα αγνοούν η μία την άλλη, δηλαδή θα είναι εχθροί. Εγώ ε, στην Ομοσπονδία ήγερα αυτό το ζήτημα και ξέρετε τι μου απάντησαν. Είναι θέμα εθνικής ταυτότητας και να μην μπλέκομαι γιατί δεν ξέρω την κατάσταση. Ε, και θα κλείσω με αυτό το σχόλιο. Ε, η παιδεία. Υπάρχει χρηματοδοτική στήριξη και για αυτά τα ζητήματα, αλλά όπως είπε η κυρία Πάκ, υπάρχουν 13 διαφορετικοί υπουργοί παιδείας. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το Tempus ε, το λένε και περισσότερο. Το Erasmus Mundus αντιμετωπίζει μεγαλύτερε δυσκολίε για του λόγου που αναφέρατε. Δεν υπήρχε εθνικό σημείο επαφή δηλαδή για να ενημερώνει τα πανεπιστήμια και το καθεξή. Ε, τώρα επιταχύνεται αλλά αντιμετωπίζει ακόμη δυσκολίε. Είναι σημαντικό να συσπηρωθούμε και να ασκήσουμε πίεση ε, για ε, ε, υπεύθυνη ηγεσία και να δώσουμε απτές αποδείξεις στους πολίτες ότι το μέλλον τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτή την πλευρά φυσικά θα είναι σημαντικό βήμα η απελευθέρωση των θεωρήσεων και ελπίζουμε ότι και το ψήφισμά σας θα συμβάλλει τα μάλα για να διαβιβάσουμε αυτό το μήνυμα, αυτά τα μηνύματα μάλλον στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ευχαριστούμε. Τώρα λοιπόν, ε, κοιτάξτε, εξαρτάται από εσά ε, αν θα περάσουμε στο επόμενο θέμα ή όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο λίγα πράγματα να πω που τα ξέχασα και εγώ. Ευχαριστώ τον Έντουαρτ για το θέμα με τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτά. Μου ξέφυγε. Κανένα πρόβλημα πρόβλημα όμως είναι στη Βοσνία Ερσεγοβίνη γιατί η ανεξαρτησία ε, είναι μονίμως αντικείμενο επιθέσεων. Δεύτερον, ο Στέλφος Βέρτζιν είπε ότι δεν προβάλλουμε αρκετά το μέλλον τη Βοσνία Ερσεγοβίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Ξαναδιαβάστε το. Εγώ νομίζω ότι προβάλλεται. Και η κυρία Κοπά, που δεν είναι πια εδώ, θα ήθελα να της πω ότι και εμένα και κανέναν άλλον στο Κοινοβούλιο δεν θα μας προσέξουν αν δεν λέμε την αλήθεια, αν δεν είμαστε ρεαλιστές. Το να είμαστε ευγενικοί, καλό είναι αυτό, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαι αγενής, απλά λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αν ακούσετε τον κύριο Ντόντικ θα καταλάβετε κι εσείς ότι και εκείνος ε, ε, καταλαβαίνει μόνο εφόσον λέει κανείς ε, τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, ευχαριστώ για την πρόταση. Και κάτι άλλο. Είπατε ότι αν υπάρχει ένας χάρτης πορείας που να είναι σαφές, τότε αυτοί θα μπορούν να εργαστούν. Δεν είναι αλήθεια. Έχουν εδώ και αρκετό καιρό χάρτη πορείας για να φύγει ο ύπατος εκπρόσωπος. Δεν έκαναν τίποτα. Αυτό όμως ε, του αφορά τους ίδιους. Τώρα στο χάρτη πορείας για την ε, ελευθέρωση ε, στις θεωρήσεις εκεί προχώρησαν για να φωλήσουν τους πολίτες στο άλλο όμως που θα χάσουν οι ίδιοι δεν το έκαναν με ρώτησαν τι πιστεύω για την πρόταση του Προεδρείου και των ΗΠΑ ψήφισμα Μαδρίτης τίποτα δεν πιστεύω γι' αυτό μπήκε απ' έξω στο παραπέντε και δεν ε, λαμβάνει υπόψη του το τι ακριβώς έχει γίνει. Το ίδιο λάθος που έκαναν πέρυσι ο κύριος Μπίλτ και οι άλλοι. Δηλαδή απ' έξω επέβαλαν κάτι αντί να πάρουν αυτό που το έχουν κάνει άλλοι. Και Επισημένω υπάρχει μια συμφωνία, η οποία βέβαια δεν εφαρμόζεται, η οποία όμως αντικατοπτρίζει το τι πιστεύουν οι πολιτικοί. Τώρα τον έρχομαι εγώ απ' έξω και να επιβάλλω τις απόψεις μου. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζω τη Βοσνία Νησοκοπίνη ως προτεκτοράτο. Ε, ό,τι άκουσα από τον Ντόντι ε, και, από άλλους... Ε, Εκτός ήταν Τζούτζικ, ε, κανείς δεν είπε ότι θέλει να υπογράψει αυτό το σχέδιο. Όσον αφορά τη διάσκεψη της 1ης ε, Ιουνίου, αυτή είναι για τη βιτρίνα. Αν θέλετε να πάτε, ας πάτε. Δεν ξέρω ποιον θα εξυπηρετήσει. Να πω για άλλη μια φορά ότι εγώ πιστεύω ότι η απαλλαγή ε, θεώρησης θα πρέπει να γίνει αυτό το καλοκαίρι. Ο συνάδελφος κ. Μιγκαρέλη είπε ότι αν ε, δώσουμε χάρτη πορείας για τη θεώρηση, τότε κάτι θα έχει εκπληρωθεί. Ε, υπάρχει η ε, ελευθέρωση και πρέπει να τους δοθούν όλα τα υπόλοιπα, όπως συνέβη και με την Αλβανία. Είπα εκπρόσωποι και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνώ με σένα. Μόνο που σε μένα δεν είναι το ερώτημα κατά πόσον ο ύπατος εκπρόσωπος ε, ε, θα είναι υπό την Lady Ashton ή κατά πόσον θα παραμείνει αντιπροσωπεία ως έχει. Αυτό ε, δεν ταιριάζει στην έκθεση, είναι εκτός. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε πράγματι, έχεις δίκιο να αναφέρουμε και τα δύο αξιώματα. Αγαπητέ κύριε Μιρέλ, έχουμε ε, συναντηθεί σε ε, συνέδρια που ήταν σημαντικότερα από αυτό της 1ης Ιουνίου. Είπατε να ε, τοποθετηθεί επιτάπητος φέτος αλλά και πέρυσι ο κύριος Μπίλτ είπανε ότι θα τοποθετήσουν, θα υποβάλουν. Έχουν την δύναμη. Για καιρό επόσαν τα πράγματα αλλά δεν γνωρίζω γιατί πιστεύουμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα καλύτερα. Και όλοι εκείνοι που είπαν ότι είναι πολύ σημαντικό να τροποποιηθεί το Σύνταγμα, συμφωνώ με αυτούς, αλλά αυτό το προσπαθούμε εδώ και καιρό να πείσουμε τους πολίτες. Εμείς δεν μπορούμε απ' έξω σε αυτή τη χώρα να επιβάλλουμε ένα νέο Σύνταγμα, εκτός αν υπάρξει μια δεύτερη συμφωνία Dayton. Εκεί έχουμε μονίμως εκλογές, έχουμε ε, υπεύθυνου πολιτικούς, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δουλέψουν μόνοι τους για το σύνταγμά τους. Ε, έλαβα υπόψη μου όλα όσα είπατε και εκεί όπου ε, μπορώ να βελτιώσω κάτι θα βελτιώσω. Πρόεδρος, ε, δεν ξέρω αν η χώρα θα ήταν σε καλύτερη μοίρα αν μιλάγαμε λιγότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπα ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί τη συζήτηση γιατί υπάρχουν ε, πάρα πολλά ε, πράγματα. Τώρα, η κυρία Νίλσεν. Να πω πρώτα ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών είναι 13 Απριλίου ε, το μεσημέρι. Και τώρα θα ήθελα να ε, καλέσω την κυρία Νίλσεν, Κιλ Νίλσεν, να αρχίσει να παρουσιάζει τη δική της την έκθεση που συστήνει ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών δεν πρέπει να δεχθεί τη συμφωνία με το Πακιστάν. Και θα ήθελα να ξέρετε και κάτι άλλο, θα σας το πω όταν τελειώσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Έχετε το σχέδιο γνωμοδότησης, το έχετε λάβει. Εκεί πράγματι συστήνω εκ μέρου τη επιτροπή μα, στην Επιτροπή Λίμπε, να απορρίψει αυτή τη συμφωνία επανεισδοχή. Και έχετε και την αιτιολόγηση τη πρότασή μου. Το επιχείρημά μου βασίζεται στα εξή δύο συμπεράσματα. Για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την ιστορική σημασία σε ευκαιρία να αξιολογεί τις συμφωνίες ε, επανεισδοχής και να επηρεάσει και το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα. Έπειτα, η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Πακιστάν ε, πρέπει να μελετηθεί περισσότερο σε βάθος. Όπως ξέρετε, οι συμφωνίες επανεισδοχής με, το, με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εγκριθεί και στο παρελθόν, χωρίς όμως να μπορεί να έχει λόγο επ' αυτών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξάλλου από τις 11 αυτές συμφωνίες δεν έχει αξιολογηθεί καμία ε, ξανά μέχρι σήμερα. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ούτε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε τα Εθνικά Κοινοβούλια. Συνεπώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λόγο ύπαρξης που ο λόγο ύπαρξή του κανονικά είναι να αξιολογεί την κοινοτική δράση και να συμμετέχει στην εκπόνηση της κοινοτικής νομοθεσία. Η αξιολόγηση αυτή για μένα είναι αναγκαία ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, πριν προχωρήσουμε στη σύναψη νέων συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποσχεθεί αξιολόγηση των συμφωνιών που ισχύουν και μάλιστα αυτό πριν από το τέλος του 2009. Δεν έχει γίνει όμως αυτό ακόμα. Συνεπώς σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση συγκρίσιμη με την κατάσταση που είχαμε με τη συμφωνία SWIFT τελικά δεν είναι τόσο η συμφωνία αυτή καθ' αυτή Ευρωπαϊκής Ένωσης με Πακιστάν, που τίθεται υπό σφισβήτηση, αλλά γενικά οι συμφωνίες ε, επανεισδοχής. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για μια πρώτη συμφωνία, και επιμένω πάνω σε αυτό, η οποία συζητιέται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τότε που άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, εφ' εξής, το Κοινοβούλιο έχει ζωτική σημασία ρόλο γιατί μπορεί να προβάλλει βέτο για τέτοιες συμφωνίες. Προτείνω λοιπόν και συστήνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει το ρόλο του που είναι ρόλος συνομοθέτη μαζί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και προτείνω να απορρίψουμε τη συμφωνία αυτή Ευρωπαϊκής Ένωσης Παϊκιστάν, ως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έχει παρουσιάσει αξιολόγηση των προηγούμενων αντίστοιχων συμφωνιών. Επίσης θέλω για άλλη μια φορά να σημειώσω ότι οι αμφιβολίες μου έχουν να κάνουν με την έλλειψη εγγύσεων όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2005 που εξηγεί για τις συμφωνίες αυτές ότι κάθε απόφαση που λαμβάνεται από τις αρμόδιες ε, αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επανεισδοχή θα πρέπει να τηρεί τη Συμφωνία τη Γενέβη του 51, το πρωτόκολλο επίσης του 67 και τη διεθνή συμφωνίες όπως είναι η Σύμβαση του Δουβλίνου του 1993 και τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 50. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και παραθέτω, κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί, να εκδιωχθεί ή να εκδοθεί από μια χώρα σε μια χώρα στην οποία κινδυνεύει με τη θανατική ποινή, με βασανισμούς ή με άλλες ε, ποινές απάνθρωπης συμπεριφοράς. Και συμφωνεί επίσης ότι στο Πακιστάν υπάρχουν παραβιάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θανατική ποινή, βασανισμοί, ε, εγκλήματα τιμή, ε, βία σε βάρος των γυναικών κλπ. κλπ. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν υπογράψει συμφωνία επανεδοχή με χώρα για την οποία δεν έχουμε καμία εγγύηση όσον αφορά την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξάλλου δεν προβλέπεται στη συμφωνία καμιά τέτοια εγγύηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το τη ρωτήσαμε, μας απάντησε ότι είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να διασφαλίζουν ότι ε, δεν θα παραβιαστούν ανθρώπινα δικαιώματα στο Πακιστάν. Δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, μη δεχτούν αυτή τη συμφωνία. Όμως, το, στο άρθρο 11 λέει ότι η θεματοφύλακα των συνδικών είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνη πρέπει να φροντίζει για τη σωστή εκτέλεση και την τήρηση του κοινοτικού δικαίου. Όμως οι διεθνείς συμφωνίες όπως ε, αυτή η συμφωνία, όπως επίσης και εγγύσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα, είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συμβούλιο από την πλευρά του λέει ότι δεν είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των συμφωνιών που υπογράφει. Ναι, αλλά πώς, εφόσον το Συμβούλιο εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη, των οποίων οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν για την επανεισδοχή. Ποιος έχει τελικά την ευθύνη. Σαν παράδειγμα, σας υπενθυμίζω ότι μια αντίστοιχη συμφωνία με το Σρι Λάνκα δημιουργήθηκε το 2004. Παρά τα σοβαρά γεγονότα που έλαβαν χώρα εκεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν ε, σταμάτησε τη συμφωνία αυτή με τους Σταμούλ, ενώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η επιστροφή ε, ατόμων εκεί αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Εξάλλου αναρωτιέμαι για την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τους Αφγανούς που η Ευρωπαϊκή Ένωση τους στέλνει στο Πακιστάν. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα άτομα αυτά τυχαίνουν καλή συμπεριφορά στο Πακιστάν και τι θα γίνει, στέλνονται μετά στο Αφγανιστάν κάτω από παράδεκτέ συνθήκε. Γιατί είναι ντόμινο η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει μια συμφωνία με το Πακιστάν και μετά το Πακιστάν υπογράφει μια συμφωνία διμερός με το Αφγανιστάν όπου δεν γνωρίζουμε ούτε ποιε είναι οι συνθήκε εφαρμογή μια τέτοια συμφωνία, ούτε καν το περιεχόμενό τη. Εξάλλου, 23 Μαρτίου, όταν το ρώτησε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα θυμόσαστε ότι δεν μου απάντησε. Εν Θέλω εδώ να αναφερθώ στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2003 που καλεί και παραθέτω τα κράτη-μέλη να τροποποιούν τους κανόνες και τις πρακτικές ε, εκδόσεων διότι και απελάσσουν γιατί πολύ συχνά γίνονται ε, την παραβάση ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και θέλω και να απαντήσω σύντομα και στους συναδέρφους που πήραν το λόγο την πρώτη φορά που συζήτησαμε αυτό το θέμα όλοι αναγνωρίσαν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τίθεται με τη συμφωνία αυτή. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι από αυτού είπαν να ψηφιστεί η συμφωνία. Είπαν ότι υπάρχουν κάποιε βελτιώσει στο Πακιστάν, χωρί όμω να μα δώσουν τα παραδείγματα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποιε είναι αυτέ οι βελτιώσει. Μα είπαν επίση ότι η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όντω είναι ευαίσθητη στη χώρα αυτή, αλλά είναι μια χώρα εταίρο στον αγώνα μα κατά τη τρομοκρατία. Και άρα πρέπει να φροντίσουμε να προχωρήσει. Σα υπενθυμίζω ότι οι συμφωνίε πληροφοριών του Πακιστάν υποστήριζαν πάντα τους Ταλιμπάν και ξεχνάνε τις ευθύνες που έχουν στο δράμα που υφίστανται οι Αφγανοί και οι Αφγανές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πρέντα και μετά ο κύριος Βιγγένη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρεις ε, παρατηρήσεις θα κάνω για την έκθεση κυρίας ε, Κινήσεν. Ε, φυσικά συμμερίζομαι την ανησυχία της κυρίας Κιλνίλσεν για την ασταθή κατάσταση που επικρατεί στο Πακιστάν, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την εσωτερική ασφάλεια. Αυτό που μόλις συνέβη τη Δευτέρα το απόγευμα, δηλαδή στο βορειοδυτικό Πακιστάν, μας δείχνει πώς χωλαίνει η κατάσταση ως προς την ασφάλεια παρακολουθήσεις της κατάστασης ε, οφείλουμε να έχουμε σαφείς όρους για τη συνεργασία για τη Συμφωνία Επανεισδοχής παρά να ε, διατρέξουμε τον κίνδυνο κάθε κράτος με τη σειρά του πέρα από ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο να βασίζεται σε αυτοσχέδιες νομικές βάσεις. βασί του άρθρου 16 της Συμφωνίας εξάλλου Υπάρχει η Μικτή Επιτροπή για την Επανεισδοχή και εκεί εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό τη επιτρέπει να παρακολουθεί αν υπάρχει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια τη επανεισδοχή. Θα έχει σαφή ρόλο έτσι η Επιτροπή. Για τους ε, Αφγανούς πρόσφυγες τώρα, λέει η κυρία Κινίλσεν ότι αν εγκριθεί η συμφωνία, τι σημαίνει αυτό αυτόματα, ε, πώς ε, ε, επαναπροωθούμε τους Αφγανούς ε, χωρίς καμία εγγύηση, χωρίς κανένα, καμία δυνατότητα έλεγχου, ελέγχου για το αν επιστρέφουν σε μια ασφαλή κατάσταση. 5 εκατομμύρια Αφγανοί επαναπατρίζονται στο Αφγανιστάν ε, σε θελούσια βάση στην πλειοψηφία των ε, περιπτώσεων υπό τη στενή υποπτία ε, της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ. Έχει ισχυρή παρουσία η τη αρμοστία σε αυτή τη χώρα και μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση των προσφύγων. Άρα και πάλι, ε, κατά τη γνώμη μου, ε, θα ήταν ευνοϊκή η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, και συμφωνώ με την κυρία Κιλ Νίλσεν, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για την εφαρμογή των ε, συμφωνιών επανεισδοχής που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εξετάσουμε εις βάθος αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν είναι αυτό επιχείρημα οπωσδήποτε για να απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να συλλέξουμε τα δεδομένα για αυτές τις συμφωνίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι επιχείρημα κατά τη σύναψη αυτής της συμφωνίας Δοχής και θα κλείσω. Thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε πολύ πολύ σύντομα, γιατί πραγματικά νομίζω δεν έχουμε πια χρόνο. Ε, σε γενικές γραμμές ε, Σημερίζομαι αυτά που είπε η κυρία Κιλ Νίλσεν δούλεψε πάρα πολύ για αυτό το σχέδιο της γνωμοδότησης. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν χώρες όπου η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι καλύτερη από ό,τι στο Πακιστάν. Και υπάρχουν τέτοιες ε, συμφωνίες επανεισδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις χώρες. Γι' αυτό λοιπόν ε, χρειαζόμαστε ε, την αξιολόγηση ε, εφαρμογής αυτής αυτών των ε, συμφωνιών επανιστοχής. Για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τις εξουσίες μας. Το θέμα δεν είναι ότι τώρα είμαστε πιο δυνατοί, αλλά έχουμε πλέον περισσότερες δυνατότητες να ζητήσουμε τέτοιου είδους αξιολόγηση και να επισημάνουμε τα θέματα που αναφέρετε και εσείς στην έκθεσή σας. Να πω το εξής. Πιστεύετε ότι μπορούμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών όχι να απορρίψει αλλά να αναβάλει αυτή την συμφωνία επανιστοχής ίσως μπορούμε να περιμένουμε πρώτα την ε, μελέτη επιπτώσεων ε, δεύτερον, ε, να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της Επιτροπής. Πώς μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι αυτή η συμφωνία επανεισδοχής θα λαμβάνει υπόψη της και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που εμπίπτουν σε αυτή τη συμφωνία επανεισδοχής. Αν λοιπόν δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αυτή η αναβολή, δεχόμεθα ως Επιτροπή αυτή τη σύσταση και εξ όσων γνωρίζω και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και αυτή ε, συζητάει το να υπάρξει ενδεχομένως το, ένα τέτοιο αποτέλεσμα της ε, ψηφορίας. Πρέπει ε, να ρωτήσω, ρωτήσω κατά πόσον είναι εδώ ο εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής. Θέλετε να μιλήσετε. Είμαι ο Πάρος ο κύριος Χάινο δεν μπορούσε να έρθει. Εγώ είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων. Μία μόνο φράση πέστε. Υπήρξαν, ετέθησαν αρκετά θέματα και θα ήθελα να απαντήσω ορισμένα από αυτά. Κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα με τους ε, διερμηνείς. Έχουν ήδη ξεπεράσει το ωράριο εργασίας τους. και θα έλεγα να το συζητήσετε απευθείας με την κυρία Νίλσεν και θα έλεγα η κυρία Νίλσεν. Μπορείτε επίσης να απαντήσετε και γραπτά. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο θέματα. Να είσαστε, αν έχετε καλοσύνη, πολύ σύντομος. Δύο θέματα αφορούν στην αρχή των ε, συμφωνιών επανιστοχής και δεύτερον στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αξιολόγηση και ημερομηνία. Εμείς ε, πρόκειται να αξιολογήσουμε ε, τις συμφωνίες επανιστοχής και αυτές που υπάρχουν και τις εντολές διαπραγμάτευσης. Όμως η καταληκτική ημερομηνία είναι το 10 και όχι το 9 και αυτή η ημερομηνία θα γίνει σεβαστή. Και έτσι φτάνω στο, στη δεύτερη παρατήρησή μου στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω να υπογραμμίσω και αυτό είναι κάτι ε, το οποίο προσπάθησα να σε επισημάνω ήδη την τελευταία φορά. Οι συμφωνίες ε, επανεισδοχής ε, δεν είναι κάτι όπου επαναλαμβάνουμε δικαιώματα που βρίσκονται κάπου αλλού. Υπάρχει μία ρήτρα και αναφέρει με απόλυτη σαφήνεια ότι η ευθύνη απορρέει από το διεθνές δίκαιο για κάθε μία από τις πλευρές και δεν ε, έρονται αυτές οι ευθύνες ε, λόγω της σύνεψης ε, μιας καινούργιας συμφωνίας. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν σεβαστά πριν περάσουμε στην εφαρμογή της συμφωνίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Κίλ Νίλσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι το Πακιστάν δεν έχει υιοθετήσει διάφορες διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμβαστής τα κτλ. Οπότε δεν με καθησυχάζεται. Αλλά θέλω να απαντήσω στον κύριο που με ρώτησε κατά πόσο μπορούμε να περιμένουμε την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, προβλέπεται για τα τέλη της χρονιάς. 2010. Που σημαίνει ότι θα αναβάλουμε, γιατί εγώ συμφωνώ να περιμένουμε την αξιολόγηση, πιστεύω ότι είναι σημαντικό, και να το ξανασυζητήσουμε τότε, αφού έχουμε την αξιολόγηση και την έχουμε μελετήσει. Αυτό συμφωνώ, απόλυτα. Αλλά δεν ήταν το μόνο που με απασχολούσε και με απασχολεί, αλλά σίγουρα θα ήταν καλύτερα να περιμένουμε την αξιολόγηση και μετά να τα ξαναπούμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, αλλά στο μεταξύ έχω να κάνω δύο-τρία σημεία. Πολύ σύντομα. Όταν ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε και για την, μόνο για την τελευταία παράγραφο που υπάρχει η σύσταση. Εάν χρειαστεί ε, να τροποποιήσουμε το κείμενο, πρέπει να γίνουν μόνο για αυτή την τελευταία σύσταση. Παρασκευή 9 Απριλίου στις 12 είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες και η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 27-28 Απριλίου και ο Πρόεδρος ευχαριστεί και πάλι στους διερμηνείς.